Bueno, Σας έδωσα πέντε λεπτά. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Παρακαλώ να καθίσετε. Και παρακαλώ να βρείτε όλοι τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας, γιατί έχουμε πάρα πολλές ψηφοφορίες και θα ήθελα να κάνετε και λίγο ησυχία για να μην αναγκάζομαι να φωνάζω κι εγώ. Πρώτο σημείο της ημερήσια. Ναι, κυρία Ρόντε, συγγνώμη, να σας δώσω το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία παράκληση. Χρειαζόμαστε... Πρέπει να διακόψουμε την ε, συνεδρίαση. Θέλω να το λάβετε υπόψη. Το έχω ξαναπεί. Πριν ε, καταλήξουμε στην καταληκτική ψηφοφορία παρακαλώ να μου δώσετε πέντε λεπτάκια, να διακόψουμε την συνεδρίαση για πέντε λεπτάκια πριν την τελική ψηφοφορία. Δεν άκουσα καλά πριν την έναρξη της ψηφοφορίας ή πριν την έναρξη της τελικής ψηφοφορίας. Πριν την τελική ψηφοφορία, Πρόεδρε. Perfecto. A ver, ¿qué es esto? No, me Υιοθετούμε λοιπόν την ημερήσια διάταξη. Εάν δεν έχετε αντιρρήσει να την εγκρίνουμε. Να εγκρίνουμε τα πρακτικά ε, των προηγούμενων συνεδριάσεων. Λοιπόν, εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσει κατά τη διάρκεια τη απογευματινή μα συνεδρίασης σήμερα και αύριο το πρωί θα θεωρηθούν εγκριθέντα τα πρακτικά. Στις 28 Οκτωβρίου θα λάβει χώρα ε, ο τριμερής διάλογος για τα εξωτικά είδη. Αυτό αποτελεί μέρο των ανακοινώσεων τη Προέδρου. Περνάμε λοιπόν ευθύ αμέσω στο σημείο 4 τη ημερήσια διάταξη. Έκθεση Γκρομπάρτσικ, τροποποίηση του κανονισμού 2187-2005 του Συμβουλίου, ως προς την απαγόρευση διαλογής αλλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας για την αλληλεία της ε, χωματίδας και του καλκανιού στη Βαλτική θάλασσα, στο Μπέλτς και στο Σούντο. Η συγητής είναι ο κ. Γκρόμπαρτσικ. Εάν δεν θέλει να παρέμβει, μπορούμε κατευθείαν να περάσουμε στη ψηφοφορία. Μήπως θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. Sorry. Ε, w zasadzie chciałbym, żebyśmy e, e, Θα ήθελα να περάσουμε στην ψηφοφορία, Πρόεδρε, αλλά να κάνω ένα σχόλιο. Ήθελα να υποβάλω μία προφορική τροπολογία που σχετίζεται με το αίτημα του Ευρωπαϊκού, ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το, να μπει ο όρος 20 δηλαδή 20η ημέρα που έχει να κάνει με την νομοθετική διαδικασία ώστε να έρθει φέτος σε ισχύ ο κανονισμός και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, σκιώδεις συζητητές ε, που με βοήθησαν. Ευχαριστώ. Καλώς. Περνούμε στην ψηφοφορία λοιπόν. Τροπολογία υπαριθμών 1 Παράγραφος 1α. Ποιος είναι υπέρ. Α, ξεκινάει η ψηφοφορία. Συγγνώμη, δεν το είπα. Σε la Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομοφόνος. Προχωρούμε στην ψήφιση της προφορικής τροπολογίας, ε, ε, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται επίσης ομοφόνος. Ψηφίζουμε την ομοθετική πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομοφόνος. Ψηφίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 22 ψήφοι υπέρ. Καμία κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται ομοφόνος η έκθεση του κυρίου Γκρόμπαρτσεκ. Συγχαρητήρια, κύριε Σιγητά. Περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Πολιετές σχέδιο για το δυτικό απόθεμα Σαφριδιού και για την αλία του αποθέματος αυτού. Εισηγητής ο κύριος Γκάλαχερ. Θα θυμάστε ότι την πρόταση αυτή την παρουσιάσαμε πριν από ένα χρόνο, χρόνο σχεδόν. Εν τω μεταξύ τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, είχαμε ψηφοφορία ανατολιστική και επειδή υπήρξε πρόβλημα με το Συμβούλιο για τα θέματα νομικής βάσης, είχαμε την πρώτη ανάγνωση για να πετύχουμε συμβαστική λύση με το Συμβούλιο. Θα θυμάστε ότι ξεκίνησε διαδικασία για την ψηφοφορία. Καλωσορίσατε ορίσατε κύριε Μάτα. Να δώσω το λόγο στο εισηγητή, μήπως θέλει να παρέμβει, αλλιώς περνούμε κατευθείαν στην ψήφιση. Έχετε το λόγο κύριε Γκάλαχερ. Ευχαριστώ. Επ' ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης συζητητές για τη συνεργασία τους και για την προσπάθειά τους να δώσουμε συνέχεια με αυτή την έκθεση, να την προχωρήσουμε. Σωστά είπατε ότι ασχολούμαστε με την έκθεση αυτή εδώ και παραπάνω από ένα χρόνο. Και φυσικά υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω της υιοθέτηση της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Δεν ήμασταν σε θέση να λάβουμε απόφαση και να ψηφίσουμε στο, στο Στρασβούργο 1η Δεκεμβρίου. Ήταν απλώς μια προσανατολιστική ψήφος αυτή. Μια προσανατολιστική ψηφοφορία. Χρειάστηκε επομένως ε, όλο αυτό το διάστημα και χάρη στον χρόνο που είχαμε να εστιάσαμε αρκετά σε αυτήν την έκθεση. Ε, και φυσικά πρέπει να χωρίσουμε και κάποιες λειτουργίες ε, στα πλαίσια Διαχειριστικής Επιτροπής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση της Προεδρίας, στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ, να δώσει στο Συμβούλιο μια ευελιξία, ούτω ώστε να καθορίσει το ελάχιστο απόθεμα αυτού του, του αλλιεύματος, Αν δεν είχαμε συμφωνήσει θα υπήρχαν δυσκολίες. Όταν συμφωνήσουν τα τρία θεσμικά όργανα, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα κάνουν καλά. Είναι το πρώτο σχέδιο διαχείρισης στα πλαίσια της συναπόφασης και είναι πολύ σημαντικό να περάσει αυτό το σχέδιο, γιατί αν δεν περάσει σωστά θα έχουμε προβλήματα και με άλλες εκθέσεις είναι μια δοκιμασία και για τις μελλοντικέ εκθέσεις. Θέλω να ευχαριστήσω την Γραμματεία της Επιτροπής Αλίας, όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου. Ε, συναντήθηκα με το Συμβούλιο κατ' επανάληψη, καθώς και το προσωπικό, την φιλελεύθερη ομάδα, τους υπαλλήλου. Θα ήθελα να πω στην Επιτροπή ότι η, η έκθεση αυτή δεν αφορά κάποιες χώρες. Ας ξεπεράσουμε τις εθνικές μας ε, διαφορές και απόψεις. Γιατί υπάρχει μια άποψη ότι μπορούμε ένα σχέδιο διαχειριστικό να το κόψουμε, ας πούμε, ε, ανάλογα με τις χώρες. Οι τροπολογίες που οδηγούν και σε συμβιβασμούς είναι να υπάρχει ένα πολιετές σχέδιο για το δυτικό απόθεμα Σαφριδιού. Υπάρχει σαφής επιστημονική συμβουλή, είναι ένα το απόθεμα και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν ενιαίο. Δεν είναι εύκολο να καθορίσουμε τα τάκα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να διαρρέσουμε το απόθεμα σε αυτό το πολιετές σχέδιο διαχείρισης. Ορισμένοι έχουν φόβους για συγκεκριμένες περιοχές. Θέλω να τους πω ότι αυτό το έχουμε λάβει υπόψη μας στην τροπολογία 20 που συνδέεται με την παράγραφο 2.1, την καινούρια. Ε, λαμβάνουμε υπόψη δηλαδή τα ιστορικά αποθέματα, τα ιστορικά ποσά. Αυτή η τροπολογία έχει γίνει αποδεκτή. Ε, συναντήθηκα στο με το Περιφερειακό Γνωμοτικό Συμβούλιο και συμφώνησε με την τροπολογία αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία υπαριθμών 19. Α, αποσύρθηκε, συγγνώμη. Τροπολογία 20 της κυρίας Αντρέ Μπαρέα. Λοιπόν, μαζί με την προφορική τροποποίηση ξεκινάει η ψηφοφορία. Se Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Αποσύρεται 21. Ε, να ψηφίσουμε τη συμβαστική λύση υπαριθμών 7. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Σε ε, τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται ομοφόνος. Προχωρούμε Στη συμβαστική λύση παριθμών 8, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. 11-11, ε, καταπίπτει, απορρίπτεται. Ναι, όταν έχουμε 11-11 απορρίπτεται. Καλώς, προχωρούμε. 22, τροπολογία 22, της κυρίας Μπιλμπάου μαζί με την προφορική ε, τροπολογία όπως τη βλέπετε. Ένρεξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. you. Ah, Απορρίπτεται. Λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 9. Έναρξη ψηφοφορίας. Σε cierra la votación. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Someto a votación la enmienda 3. Ε, πάμε τώρα στην 3. Έναρξη ψηφοφορίας. Se cierra la votación. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε από κοινού το 11... Α, τη συμβαστική λύση 11. Έναρξη ψηφοφορίας μόνο. Σε cierra la votación. Ε, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομοφόνος. Ε, το 12 τώρα παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Σε φύρρα. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Από κοινού τώρα. 13, 14, 15 και 16. Συμβαστικές τροπολογίες από κοινού ψηφίζουμε μαζί. Ε, ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται όλα. Η τέσσερα καταπίπτει για την πέντε. Ε, ψηφίζουμε την τροπολογία υπαριθμών πέντε. Ξεκινούμε. Ε, πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Αποσύρθηκε η 6 Πάμε στην 25. Έναρξη ψηφοφορίας. Σε θύρα λαβοτσαφίαν. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται ομοφόνος. Ψηφίζουμε το δεύτερο μέρος της τροπολογίας υπαριθμών 24. Έναρξη ψηφοφορίας. Σε θύρα Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 14 κατά 9 υπέρ. la enmienda νούμερο 7. Ψηφίζουμε την 7. Έναρξη ψηφοφορίας. Se cierra la votación. Adoptado. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε από κοινού τις συμβαστικές τροπολογίες 17 και 18. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνονται ομοφόνος. Καταπίπτει η τροπολογία υπαριθμών 8 και ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 19. Έναρξη ψηφοφορίας. Σε Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται, άρα καταπίπτει η 9. Ψηφίζουμε την 20, του τροπολογίου υπαριθμών 20. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Mm, εγκρίνεται. Αποσύρθηκαν οι 10 και οι 26. Ψηφίζουμε την συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 21. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Αποσύρεται, έχει αποσυρθεί 11 και 27. Ψηφίζουμε επομένως την τροπολογία υπαριθμών 12. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Αποσύρθηκε 28. Ψηφίζουμε την τροπολογία 13. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Λοιπόν, ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 22, έναρξη της ψηφοφορίας. Σε θύρα. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Αποσύρθηκε η 29. Ψηφίζουμε τώρα τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1 και την συμβαστική λύση υπαριθμών 3. Από κοινού και τις δύο. Ψηφίζουμε. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Εγκρίνονται μαζί. Ψηφίζουμε την 2. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 2. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Αποσύρθηκε η, η τροπολογία 1 και η 14. Η 15 καταπίπτει από τη στιγμή που έγιναν δεκτές οι προηγούμενες συμβαστικές τροπολογίες. Ψηφίζουμε την 4, συμβαστική τροπολογία 4. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται ομοφόνος. Τροπολογία υπαριθμών 2 του εισηγητή. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομοφόνος. 16 της κυρίας Αντρές Μπαρέα. Συμβατεί με την 2 του εισηγητή μαζί με την προφορική τροπολογία που βλέπετε στο κείμενο. Έναρξη της ψηφοφορίας. Σε la votación. Aprobada. Eh, Εγκρίνεται. Άρα η συμβαστική η τροπολογία υπαριθμών 5 καταπίπτει. Εάν δεν κάνω λάθος, επιτρέψτε μου να το ελέγξω. Εγκρίθηκαν οι συμβαστικές τροπολογίες 13, 14 και 15. Όχι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ε, ε, ψηφίζουμε τη συμβαστική λύση υπαριθμών 5. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέραστη της ψηφοφορίας. Άρα εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει. Επομένως, καταπίπτει ή όχι. Καταπίπτει, ναι. Ψηφίζουμε την 18. Α, καταπίπτει και η 18. Επομένως, αφού μου ζήτησε η κυρία Ρόντος, η οποία δεν με ακούει βεβαίως, αφού μου ζήτησε λοιπόν να διακόψουμε την ψηφορία και να της δώσουμε το λόγο, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, δεν χρειάζεται για το σημείο αυτό πια να διακόψουμε. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο για ψηφοφορία. Καλώς, μήπως ε, θέλει κάποια άλλη πολιτική ομάδα να πάρει το λόγο. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν το σχέδιο νομοθετικής πρότασης όπως τροποποιήθηκε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρα της ψηφοφορίας. 22 υπέρ και μία αποχή. Συγχαρητήρια. θα εξεταστεί στη δεύτερη ολομέλεια του Νοεμβρίου. Προχωρούμε στην επόμενη έκθεση για το Γάβρο. Μακροπρόθεσμο σχέδιο για το απόθεμα γάβρου στο βισκαϊκό κόλπο. Η κυρία Μπιλμπάο είναι η συγγήτρια. Εδώ και ένα χρόνο ασχολούμαστε με την έκθεση αυτή. Το ίδιο ισχύει όπως και με την έκθεση του κυρίου Γκάλαχερ. Εν τω μεταξύ τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Είχαμε ψηφοφορία προσανατολιστική. Έγινε πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο και ούτω καθεξής. Ε, είναι γνωστά. Να δώσω το λόγο στην κυρία Μπιλμπάου πριν ε, περάσουμε στη ψηφοφορία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να πω πολύ απλά ότι σκοπός του μακροπρόθεσμου αυτού του σχεδίου διαχείρισης ήταν να δοθεί περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη αυστηρότητα, αν θέλετε, περισσότερη επιστημονική ακαμψία στη διαχείριση του θέματος, σύμφωνα με τις ε, γνωμοδοτήσεις τις επιστημονικές. Δηλαδή να βγαίνει αυτόματα το συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα. Γνωρίζετε όλη τη διαδρομή που έχουμε ακολουθήσει με αρκετά εμπόδια. Θα είναι περίεργη η ψηφοφορία σήμερα. Το Συμβούλιο ζήτησε από την Επίτροπο να αποσύρει το μακροπρόθεσμο αυτό σχέδιο. Το γνωρίζουμε αυτό. Και μέχρι την περασμένη εβδομάδα που είχαμε συναντηθεί με την Επίτροπο, μας είχε πει ότι δεν ήξερε ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Θα ήθελα να πω ότι το σχέδιο αυτό θα εφαρμοστεί σε ένα συγκεκριμένο κλάδο, και το υπογραμμίζω αυτό, έναν κλάδο πάρα πολύ υπεύθυνο και έχει αποδείξει την υπευθυνότητά του αυτή, έχει ακολουθήσει πρακτικές πολύ καλές τον τελευταίο καιρό και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την υπευθυνότητα του κλάδου. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να τονίσω το εξή. Να λάβετε υπόψη σα τα επιχειρήματα που είχαμε με όλε τι κοινοβουλευτικέ ομάδε, να λάβετε υπόψη την επιχειρηματολογία για το 0,4% για τη συμβαστική τροπολογία 6 για την 11 σε περίπτωση απουσίας πληροφόρησης να μην έχουμε μείωση ε, κάτω του 10% και να μην πέσει το ΤΑΚ κάτω από τους 7.000 τόνους, το συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα, διότι δεν φταίει ο κλάδος αν έχουμε αποσία ή Δεν είναι δίκαιο να τιμωρήσουμε τον κλάδο για τους λόγους αυτούς. Και, κυρία Πρόεδρε, στη Συμβαστική Τροπολογία Παριθμών 24, ως προς το περιθώριο ανοχής και σήμερα και το πρωί και στο παρελθόν, έχω μιλήσει με διαφόρους βουλευτές θα ήθελα λοιπόν αυτό το περιθώριο ανοχής να είναι της τάξης του 10%. Η Επιτροπή επιθυμούσε το 5%, όμως το Δεκέμβριο ενέκρινε 20%. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα να είναι στο 10% αυτό το περιθώριο. Καλώς. Λέει η Πρόεδρος, προχωρούμε στη ψηφοφορία. Η 23 αποσύρθηκε. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 6. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 13 ψήφοι κατά, 9 υπέρ. Απορρίπτεται η 6. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 7. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται η 3 καταπίπτει, η 4 αποσύρθηκε. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 8. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 9. Συμβαστική τροπολογία 9. Έναρξη της ψηφοφορίας. Se cierra la votación. Aprobado. Eh, Πέρα της προφορίας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 27. Έναρξη της προφορίας. Se cierra la votación. Πέρα της προφορίας απορρίπτεται. El compromiso número 10. Se abre la votación. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 10. Έναρξη της προφορίας. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 11. Έναρξη της ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται 12 κατά 10 υπέρ. Ψηφίζουμε την 29. Έναρξη της ψηφοφορίας. Se cierra la Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 13 κατά, 9 υπέρ. Ψηφίζουμε την 28. Έναρξη ψηφοφορία. Se cierra la votación. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Την 31 ψηφίζουμε. Έναρξη ψηφοφορία. Σε cierra la votación. Πέραση τη ψηφοφορία. Rechazada. Someto a votación la enmienda número 30. Se abre la votación. Ε, ψηφίζουμε την 30. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται επίσης. 12 κατά 10 υπέρ. Η 5 αποσύρθηκε. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 12. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το άρθρο 6 και τις συμβαστικές τροπολογίες 13, 14 και 15 μαζί. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Ψηφίζουμε το άρθρο 7, έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 16 επίσης ε, προσαρμογή του κανονισμού ελέγχου. Έναρξη ψηφοφορίας. Σε cierra la Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται. Το άρθρο 10, το οποίο είναι το ίδιο. Έναρξη ψηφοφορίας. Se cierra. Aprobado. Somete a votación el compromiso. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 17. Έναρξη ψηφοφορίας. Σε θύρα. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται 17 υπέρ 5 κατά. Εάν συμφωνείτε να ψηφίσουμε ε, τα τρία επόμενα άρθρα μαζί. 11.2, 11.3 και 12. Ψηφίζουμε από κοινού τα τρία αυτά άρθρα ε, που είναι κανονισμός ελέγχου προσαρμογής. Έναρξη ψηφοφορίας, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνονται, ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμό 18, έναρξη της ψηφοφορίας. Σε θύρα. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Επομένως, καταπίπτει η τροπολογία 33, αλλά και η τροπολογία υπαριθμών 7. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 19. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 13 υπέρ, 9 κατά, 13 υπέρ. Επομένως καταπίπτει η 34 αλλά και η 8. Ψηφίζουμε τις συμβαστικές τροπολογίες 20 και 21 μαζί. Σε la votación. Πέρας της ψηφοφορίας. Επομένως καταπίπτει η 9. Ψηφίζουμε τον κανονισμό ελέγχου προσαρμογής ως προς το άρθρο 14. Έναρξη της ψηφοφορίας. Παράγραφος 3. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική λύση παριθμών 22. Πέρας της ψηφοφορίας ψηφίζουμε την 23. Πέρας της ψηφοφορίας Ψηφίζουμε το άρθρο 15.3, κανονισμός ελέγχου προσαρμογής, έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε τη συμβαστική λύση υπαριθμών 24 μαζί με την προφορική τροπολογία της εισηγήτριας, δηλαδή το περιθώριο ανοχής από 20 να πάει στο 10%. Επιμένω για αυτή την προφορική τροπολογία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Επομένως, Καταπίπτει η 11, η 36, η 37. Επίσης ψηφίζουμε την 38. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το άρθρο 18. Κανονισμός ελέγχου προσαρμογής. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει επομένω η 39. Ψηφίζουμε το άρθρο 19, πρώτη παράγραφος κανονισμός ελέγχου προσαρμογής. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική λύση παριθμών 25 έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 13 ψήφοι υπέρ, 9 κατά. Επομένως καταπίπτει η τροπολογία υπαριθμών 12, γι' αυτό και ψηφίζουμε την συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 26. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 17 υπέρ, 5 κατά. Ψηφίζουμε το άρθρο 20. Κανονισμός ελέγχου προσαρμογής. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 27. Πέρας της ε, ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει επομένω η τροπολογία 14, γι' αυτό και ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 28. Πέρα της ψηφοφορία. εγκρίνεται. Επομένω, καταπίπτει η 40. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 29. Πέρα της ψηφοφορία. Εγκρίνεται 17 υπέρ 5 κατά. Ψηφίζουμε την 16. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 15 κατά, 7 υπέρ. Ψηφίζουμε την 30, συμβαστική τροπολογία 30. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται 12 ψήφοι κατά 10 υπέρ. Ψηφίζουμε την τροπολογία 41. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 21 ψήφοι κατά, 1 ψήφος υπέρ. Ψηφίζουμε Την 18. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 19 αποσύρθηκε. Αιτιολογική σκέψη υπαριθμό 4. Νομική προσαρμογή. Ψηφίζουμε αυτό. Έναρξη της ψηφοφορίας. Αιτιολογική σκέψη παριθμών 4. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 4. Ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 12 ψήφοι κατά, 10 υπέρ. Αιτιολογική σκέψη υπαριθμών 7 την ψηφίζουμε. Είναι πάλι νομική προσαρμογή. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 5 τώρα ψηφίζουμε. πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Η τροπολογία 1 αποσύρθηκε, η 21 καταπίπτει. Ψηφίζουμε την αιτιολογική σκέψη υπαριθμών 8 και ανονισμός ελέγχου προσαρμογής. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και μου ζήτησε η σοσιαλιστική ομάδα

Kelda. Yeah. prochain A ver, eh, pido, pido que, que, se, que se sienten. Παρακαλώ να καθίσετε. για να περάσουμε στην τελική ψηφοφορία. Λοιπόν, ψηφίζουμε την νομοθετική πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Έναρξη της ψηφοφορίας. Σε cierra la votación. Aprobada Πέρας της ψηφοφορίας, 13 ψήφοι υπέρ, 9 κατά. Ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας με την ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται 13 ψήφοι υπέρ 9 κατά. Buena y buena suerte. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Δεν είναι πολύ ικανοποιημένη η κυρία Μπιλμπάου, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να συγχαρούμε ε, τον εισηγητή κάθε φορά για τη δουλειά που έχει κάνει. Περνούμε τώρα στο σημείο 7. Ενδιάμεση Συμφωνία εταιρική Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κράτη, και κρατών του Ειρηνικού. Εγώ είμαι η συγκήτρια, όπως γνωρίζετε. Είναι μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου βάσει της συμφωνίας που είχαμε με τα νησιά Φίτσι, την Παππούα Νέα Γουινέα. Έχουμε μια τροπολογία της κυρίας Λεβάου και ήθελα να σας πω το εξής. Δεν είμαι κατά της τροπολογίας αυτής. Θα ήθελα όμως να σε εξεξηγήσω γιατί προτιμώ να διατηρηθεί το δικό μου κείμενο, η δική μου διατύπωση. Είναι πιο περιοριστικό, αν θέλετε, το δικό μου κείμενο. Ε, πιο περιοριστική η δική μου διατύπωση. Η ότι η πρόταση έχει προτείνει μια σειρά συνθήκων και προϋποθέσεων. Όμως, θεωρούμε ότι από αλλιευτικής σκοπιάς δεν είναι καλό πράγμα να έχουμε συνολική παρέκκληση ε, των κανονισμών για την προέλευση. Επομένως, γι' αυτό καταρχήν είμαστε αντίθετοι. Αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα. Από εκεί και πέρα, οι όροι, οι προϋποθέσεις που προτείνει η κυρία Λαβάν έχουν ως εξής. Η έκθεση προβλέπεται στο πρωτόκολλο στην ενδιάμεση αναθεώρηση των κανόνων για την προέλευση Προβλέπονται εκεί δηλαδή οι εκθέσεις αξιολόγησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς λειτουργήσε η παρέκκληση ή πώς δεν λειτουργήσε και σύν της άλλης θέλω να σας ξεκαθαρίσω το εξής. Το περιβαλλοντικό ζήτημα που είναι, είναι μία από τις προϋποθέσεις που θέτει η κυρία Λοβάουν και ουσιαστικά αποτελεί καταστροφή για τους κανόνες προέλευσης, θέλω να ξέρετε το εξής. Η ίδια η κυβέρνηση της Παππούας Νέας Γουινέας έχει θεσμοθετήσει παρεκκλήσεις από τη δική της περιβαλλοντική νομοθεσία. Επομένως, καταστάσεις που και εκχωρήσεις αν θέλετε, για να έχουμε αποθέματα, δεν μπορούν να κατοχυρηθούν ε, εκτός και αν προσφύγει κανείς στα δικαστήρια. Αυτή είναι η τροποποίηση που έχει ήδη εγκριθεί ως προς την περιβαλλοντική νομοθεσία. Δηλαδή, μία από τις προϋποθέσεις τις οποίες ζητάτε εσείς δεν τηρείται ήδη και δεν εφαρμόζεται ήδη γιατί έχουν ήδη αλλάξει τα πράγματα σε μία από αυτές τις χώρες. Και βεβαίως αν προσφύγει κανείς και στα δικαστήρια ε, θα ε, αποκτήσει δημοσιότητα το θέμα πολύ αρνητική. Από εκεί και πέρα έχουμε αγγελίες από πλευράς ε, κυβέρνησης της Παππούας Νέας Γουινέας για να, να προσελκύσουν εταιρεία, εταιρείες που ε, παρασκευάζουν κονσέρβες, η κονσερβοβιομηχανία δηλαδή. Η ίδια η κυβέρνηση του κράτους αυτού ε, διαφημίζει ελαστικές ε, εργασιακές συνθήκες, ένα πολύ ελαστικές συνθήκες ε, κοινωνική ασφάλεια ακριβώς για να προσελκύσει ε, τις εταιρείε. Από δεν έχει κανένα νόημα για να μιλούμε για αυτό το πράγμα πλέον. Και το τρίτο επιχείρημα είναι το εξής. Γίνεται λόγος για την τήρηση των ε, κανονισμών της περιφερειακής οργάνωσης αλίας για το νοτιοδυτικό ειρηνικό. Εάν πάτε στην ιστοσελίδα του περιφερειακού αυτού οργανισμού, θα αντιληφθείτε ότι τα περισσότερα από αυτά τα κράτη δεν εφαρμόζουν αυτούς τους κανονισμούς, δεν τους στηρούν και ειδικότερα οι χώρες που ουσιαστικά έχουν εταιρείε που εδρεύουν στην παπούα Νέα Γουινέα. Και έχουμε και μια ιστορία αληθινή, η οποία είναι και λίγο μακάβρια και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Εξαφανίστηκε τις προάλλες ένας παρατηρητής από την Περιφερειακή Οργάνωση Αλίας, εξαφανίστηκε ο οποίος παρατηρούσε εκφορτώσεις ε, από, και μεταφορτώσεις από σκάφη με σημαία των Φιλιππινών. Πολλά γίνονται σε αυτά τα νερά. Επομένως, είναι πιο περιοριστική η γνωμοδότηση έτσι όπως την προτείνει η εισηγήτρια. Και γι' αυτό δίνω αυτές τις εξηγήσεις δημόσια. Δεν είμαι κατά της διατύπωσης της κυρίας Λαμπάου, όμως ε, με την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, η δική μου διατύπωση είναι πιο αυστηρή, πιο άκαμπτη, πιο, πιο περιοριστική. Ε, Βεβαίω προτιμήσετε ε, την άλλη πρόταση, δεν είναι τραγωδία, θα συμφωνήσω. Η κυρία Ρόντοστ. Ξέρω ότι καθυστερώ σήμερα χωρίς να υπάρχει λόγο στην ε, συνεδρίαση, αλλά ήταν πολύ πιστικά τα επιχειρήματά σας. Ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε. Πρέπει να διακόψουμε. Φέρατε στο τραπέζι κάποια επιχειρήματα τα οποία δεν τα έχουμε συζητήσει. Κοιτάξτε, πολλά επιχειρήματα έχουν προβληθεί και στο παρελθόν. Εγώ προσπάθησα τώρα να δώσω συγκεκριμένε εξηγήσει γιατί αντιτίθεμαι σε αυτέ τι τροπολογίε, οι οποίε είναι αποδεκτέ και είναι απολύτως εύλογε και λογικέ. Αντιτίθεμαι όχι γιατί διαφωνώ επί τη ουσία, αλλά διότι θεωρώ ότι η δική μου διατύπωση κάνει το, το κείμενο πολύ πιο περιοριστικό, πολύ πιο αυστηρό. Λοιπόν, εάν θέλετε να σας δώσω ε, πέντε λεπτά, παρακαλώ. Ε, ε, ε, λοιπόν, προχωρούμε. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία της κυρίας Λοβό, έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πέντε αποχές και δύο ψήφοι υπέρ. Ψηφίζουμε τώρα το κείμενο ε, της γνωμοδότησης, του σχεδίου γνωμοδότησης, έναρξη της ψηφοφορίας. Σε φύρα. Πέρας της ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 2 κατά. Σας ευχαριστώ. Περνούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ε, έκθεση του κυρίου Γκάλαχερ. Στις 9 Νοεμβρίου του 2010 θα λάβει χώρα η ψηφοφορία στην Επιτροπή Ίντα και μετά θα περάσει στην Ολομέλεια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισλανδίας, Λίχτενστάιν και Νορβηγίας για τον χρηματοδοτικό και χρηματοοικονομικό μηχανισμό για την προγραμματική περίοδο 2009-2014 και τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένων αλλιευμάτων και αλλιευτικών προϊόντων για την ίδια περίοδο. Μήπως θα ήθελε ο εισηγητής να πάρει το λόγο σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει καμία τροπολογία. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Καλώς. Ξεκινούμε την ψηφοφορία για την έκθεση του κυρίου Γκάλαχερ. Πέρα της ψηφοφορίας. Συγχαρητήρια, κύριε Σιγητά. Εγκρίνεται ομοφόμνος. 21 ψήφοι υπέρ, καμία αποχή και καμία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Περνούμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Λήξη λοιπόν των ψηφοφοριών και τώρα τροποποίηση του κανονισμού 861 κάθετος 2006 του Συμβουλίου της 22ης Μαΐου του 2006 για τη θέσπιση κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινή αλλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του δικαίου της θάλασσας. Θα ξέρετε ότι η κοινή αλλιευτική πολιτική χρηματοδοτείται μέσα από δύο κανονισμούς. Ο ένας είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας και ο κάθε κλάδος ουσιαστικά ε, χρηματοδοτεί διαφορετικά μέτρα. Έχουμε λοιπόν την έκθεση του κυρίου Φερέιρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει πρόταση. Να δώσω το λόγο στον κύριο Φερέιρα. Να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση τροποποίησης ε, του κανονισμού 861 κάθετος 2006 παρουσιάστηκε ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε προηγούμενη συνεδρίαση. Επομένως δεν έχει νόημα να μακρηγορήσω για αυτό το σημείο. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για ένα σημαντικό χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αλία μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας. Αυτά είναι τα δύο βασικά μέσα, τα δύο βασικά εργαλεία για την ενεργοποίηση και εφαρμογή της ε, πολιτικής αλίας. Αυτός ο κανονισμός, πιο συγκεκριμένα, αφορά τους τομείς της διακυβέρνησης, των διεθνών σχέσεων. Σας παρακαλώ, ε, λέει η Πρόεδρος, ακούω πάρα πολύ θόρυβο από την Ισπανική καμπίνα. Μήπως μπορείτε να το ρυθμίσετε παρακαλώ. Ωραία, ο εισηγητής ξανά. Αυτός ο κανονισμός ε, προβλέπει τη χρηματοδότηση μέτρων στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων, του governance, της διακυβέρνησης, της συλλογής δεδομένων και επιστημονικών στοιχείων και τον έλεγχο της εφαρμογής της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως σας είπα, ήδη παρουσίασε την πρότασή της στην ε, δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή, επομένω δεν θα μακρηγορήσω επί της πρότασης αυτής. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι θεωρώ ότι οι λόγοι για τους οποίους έγινε τροποποίηση του κανονισμού είναι δικαιολογημένοι και βάσιμοι. Οι προτάσεις που παρουσιάζει η Κομισιόν, επομένως, είναι απόλυτα δικαιολογημένες. Και είναι και προσαρμοσμένες στους στόχους. Δηλαδή, να προσαρμόσουμε τον κανονισμό στη σχετική νομοθεσία. Κάποιες δράσεις χρηματοδοτούνται με περισσότερα χρήματα γιατί έχουν διευρυνθεί. Επίσης, ως συνήθως, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε κάποιες διατάξεις του καονισμού, ούτως ώστε να υλοποιήσουμε καλύτερα τις, τα μέτρα που είναι απαραίτητα. Τώρα, εγώ θέλησα να παρουσιάσω κάποιες τροπολογίες σε αυτή την ε, πρόταση τροποποίηση του κανονισμού τροπολογίε που μπορούν να μας βοηθήσουν για να ευθυγραμμίσουμε καλύτερα το νομοθέτημα αυτό, τον κανονισμό αυτό, με τις εξελίξεις του τομέα. Κυρίω θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο τροπολογίε και μετά θα μιλήσω και για μία τρίτη, τελευταία όμως. Σήμερα όλοι αναγνωρίζουν το πόσο σημαντικό είναι το να διαχειριστούμε την αλία με βάση κάποια επιστημονικά στοιχεία και κάποιες επιστημονικές γνώσεις, ε, ιδίως για το, την κατάσταση των αλλιευμάτων. Αυτή είναι μια προϋπόθεση για μια βιώσιμη εξέλιξη της αλληλευτικής δραστηριότητας. Στην έκθεση παρουσιάζεται η δυνατότητα αύξησης του βαθμού συγχρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τη συλλογή, διαχείριση και διάδοση δεδομένων. Σήμερα προβλέπουμε τη συγχρηματοδότηση του 50, σε ύψος 50% και ζητάμε να ανεβάσουμε αυτό το, ποσο, αυτό το ποσοστό και να φτάσει στα, στο 75%. Εδώ μιλάω για οικονομικές πληροφορίες, για τον αλληλευτικό στόλο, για την δατοκαλλιέργεια, για τον, για τον κλάδο εν γέννη. Εδώ θέλω να εντάξω και το περιβάλλον όλες, όλα αυτά τα δεδομένα, για αυτά τα στοιχεία που σας προανέφερα, όλη η συλλογή των δεδομένων για τα στοιχεία που σας προανέφερα, είναι απαραίτητη και επιπλέον πρέπει να συγκεντρώσουμε και πολύ περισσότερες πληροφορίες πέρα από την στατιστική ανάλυση που κάνει κάθε κράτος μέλος. Εδώ ζητούμε περισσότερες πληροφορίες και μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να βρούμε αυτές τις πληροφορίες. Επίσης υπάρχει μια απέτηση για περιφερειακές τράπεζες δεδομένων, με δυνατότητα να έχουν πρόσβαση όλα τα κράτη-μέλη τα οποία ενδιαφέρονται για μια συγκεκριμένη περιοχή, Φέρπιν, Μεσόγειος, Βόρειος Κλαντικός κτλ. Αυτή η ανάγκη αναγνωρίζεται από όλους. Όμως αυτό συνεπιφέρει μεγαλύτερες ε, επενδύσεις και μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, θα πρέπει να επιτρέψουμε ένα υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης, υψηλότερο από το 50% που είναι το σημερινό ποσοστό, αυτό που προβλέπεται δηλαδή από τον σημερινό κανονισμό. Σε ό,τι αφορά την περαιτέρω συλλογή δεδομένων, για τα οποία προτείνω την ίδια τροπολογία, δηλαδή αύξηση του βαθμού συγχρηματοδότησης ε, στο ύψος του 75%, μια και πρόκειται για έξοδα, για δράσεις ε, που προωθούνται μετά από την παρουσίαση προτάσεων, δηλαδή διαγωνισμών κτλ. Αυτό αποτελεί κίνητρο για την παρουσίαση αυτών των προγραμμάτων με σκοπό ας πούμε την προώθηση των διαγωνισμών. Αυτά για τη συλλογή δεδομένων. Τώρα, για τον έλεγχο προτείνουμε την ίδια αλλαγή, όπως δηλαδή για τη συλλογή και διαχείριση των δεδομένων και για τον έλεγχο, και για τον έλεγχο συνειδητοποιούμε ότι θα πρέπει να καταστήσουμε πιο βιώσιμο τον κλάδο. Και εδώ τα κράτη-μέλη ε, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες ανάγκες σε ό,τι αφορά την εκτέλεση της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Αυτό το συζητήσαμε και στην τελευταία ολομέλεια. Επίσης μεγαλύτερες, ε, υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσει που βαραίνουν τα κράτη-μέλη λόγω των διεθνών συμφωνιών. Έχουν ευθύνε τα κράτη-μέλη. Μεγαλύτερες ευθύνε σε επίπεδο ελέγχων λόγω διεθνών συμφωνιών. Αλλά αυτές οι μεγαλύτερες ευθύνες επισύρουν την ανάγκη συγχρηματοδότησης σε υψηλότερο ποσοστό. Όπως ακριβώς εξήγησα για τη συλλογή των δεδομένων. Αντί λοιπόν για 50% συγχρηματοδότηση για τον έλεγχο προτείνω και εδώ συγχρηματοδότηση ύψους 75%. 75% λοιπόν. Τώρα υπάρχει μια ακόμα τροπολογία που αφορά το σημερινό άρθρο 8 του κανονισμού όπου περιγράφονται τα διάφορα μέτρα και οι διάφορες δράσεις δράσεις που μπορούν να ενταχθούν στα χρηματοδοτικά μέτρα. Συμφωνώ με τα όσα είπε η Επιτροπή. Απλώς η αγορά τεχνολογίας και η εγκατάσταση του μηχανισμού για την μετάδοση των δεδομένων αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα προσθέσουμε. Όχι μόνο αγορά αλλά και ανάπτυξη τεχνολογίας ε, από μέρους των αρμοδίων εθνικών αρχών. Αυτό θέλω να το προσθέσουμε. Αυτό λέει η τροπολογία. Ακόμα τώρα μια τροπολογία στα πλαίσια της υδατοκαλλιέργειας. Εκεί μιλάμε για την συλλογή κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων. Αυτό προτείνει η Κομισιόν. Εγώ θέλω να προσθέσουμε τη δυνατότητα συλλογής περιβαλλοντικών επίσης δεδομένων δεδομένης της δυνατότητα ανάπτυξης αυτής της ε, δραστηριότητας, της υδατοκαλλιέργειας ενώ, η περιβαλλοντική διάσταση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πολύ περισσότερο. Και εξάλλου και αυτό αντανακλά και την συζήτηση που είχαμε σε αυτό εδώ το χώρο όταν μιλήσαμε για την έκθεση Μιλάνα. Σε ευθεία γραμμή μετά όσα είπαμε ξεκίνη την έκθεση και για να ενδυναμώσουμε τον, ε, τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας πρέπει λοιπόν να συλλέγουμε ε, στοιχεία και για την υδατοκαλλιέργεια. Αυτό το τελευταίο, ε, αυτή είναι η τελευταία τροπολογία μαζί με τις τροπολογίες που σας προανέφερα. Ο επόμενος ομιλητής, ευχαριστώ Πρόεδρε. Α, δεν είχα ακούσει το όνομά μου. Ε, ευχαριστώ τον εισηγητή για την ε, προσπάθειά του. Νομίζω ότι οι τροπολογίες της ε, Επιτροπής στον κανονισμό του 2006 πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Το πλαίσιο το εφαρμοστικό διευρύνθηκε, συλλογή δεδομένων από τα κράτη-μέλη, διαχείρισή τους και χρήση των δεδομένων αυτών. Καλό είναι αυτό. Τώρα, η οικονομική υποστήριξη του Συμβουλευτικού Συνεδρίου, ε, Συμβουλίου ε, διευρύνθηκε και ε, υπάρχει περιορισμός μόνο στην αρχική φάση. Επίσης προβλέπονται κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία στη συλλογή των δεδομένων. Θετικό είναι αυτό. Ο κύριος Φερέιρα όμως θέλει να αυξήσει και το Ποσοστό συγχρηματοδότηση για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση των δεδομένων από το 50% στο 75%. Λίγο επικίνδυνο μου φαίνεται αυτό, γιατί η Κομισιόν τότε νομίζω δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει τόσα πολλά προγράμματα. Σήμερα υπάρχουν ζώνες ανάπτυξη κατά προτεραιότητα και νομίζω ότι με μια τέτοια αύξηση ε, θα υπάρξει πρόβλημα. Η ισορροπία που έχουμε πετύχει με τη σημερινή κατάσταση είναι ικανοποιητική σε ό,τι αφορά το ποσοστό συγχρηματοδότηση αν φτάσουμε... Επίσης μπορούμε να πάμε στο 80% για τους τομείς κατά προτεραιότητα και η συγχρηματοδότηση είναι στο 50% για τους τομείς που δεν αποτελούν προτεραιότητα. Αν αυξήσουμε το 50% σε 75% για τομείς που δεν αποτελούν προτεραιότητα, νομίζω ότι ε, θα έχει σαν αποτέλεσμα να μειώσει την ευελιξία μας. Ευχαριστώ, κυρία Ρόντοστ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε προβλήματα με τη γερμανική μετάφραση. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε απόλυτα την ε, έκθεση και κυρίως την τροπολογία 8. Ε, δεν ξέρω μήπως μπορείτε εσείς με κάποιο τρόπο να παρέμβετε για να λαμβάνουμε καλύτερες μεταφράσεις. Ε, το έχω ξαναπεί. Τώρα για την έκθεση να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή. Πρέπει να πω εδώ ότι όπως και στις προηγούμενες συζητήσεις έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την ενίσχυση της ε, συγχρηματοδότησης. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη, μεγαλύτερος και περισσότερος έλεγχος, αλλά λιγότερος, ε, γιατί όλα τα κράτη-μέλη ε, θα ζητήσουν 75% μετά χρηματοδότηση και να δίνουν μόνο το 25% τα ίδια και οι πλούσιες χώρες θα κάνουν το ίδιο με τις, ε, πιο, με τις ε, φτωχές. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε λιγότερους ε, ελέγχους και λιγότερα δεδομένα. Δεν θα μπορέσουμε λοιπόν αυτό να το υποστηρίξουμε και θα παραμείνουμε στην άποψη που λέει ότι πρέπει αυτά να παραμείνουν στο 50%. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ρόντουστ. Σημειώνω αυτό που είπατε για τη μετάφραση. Να δώσω το λόγο στην κυρία Λόβιν. Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Φερέιρα και θα ήθελα να συμφωνήσω και με αυτά που είπε η κυρία Ρόντους για τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο από το 50% στο 75% δεν νομίζω ότι αυτό θα μας οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα, γιατί έτσι θα καλύπτονται πολύ λιγότερα προγράμματα. Ήδη υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις ε, για συγκεκριμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα, αν θέλει κανεί να επενδύσει σε αεροσκαφή ή κάποια άλλα ε, μηχανήματα τεχνολογία, νομίζω ότι αυτά παραμένουν ε, σε, είναι σε εξαίρεση. Ε, νομίζω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να αυξηθεί το επίπεδο χρηματοδότηση στο 75%. Ευχαριστώ. Uh, Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Να πω ότι εμεί στην ομάδα μα έχουμε κάποιε επιφυλάξει για την αύξηση του 50 σε 75%. Αυτό ήθελα απλώ να πω. Θα μπω σε λεπτομέρειε όταν θα μπούμε και στην ουσία του πράγματο. Ευχαριστώ. Καλώς. Λοιπόν, έχω και εγώ κάποια σχόλια. Στο άρθρο 9 μιλάτε για συγκέντρωση περιβαλλοντικών στοιχείων ή δεδομένων. Προσωπική μου άποψη είναι ότι τα περιβαλλοντικά στοιχεία πρέπει να γίνονται αντικείμενο διαχείρισης χρησιμοποιώντας την πολιτική για το περιβάλλον. Έτσι δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει στο 1 β να περιλάβουμε την αναφορά στα περιβαλλοντικά στοιχεία, εκεί όπου μιλούμε για τα συμπληρωματικά στοιχεία. Εάν συμφωνείτε, πιστεύω ότι αυτό είναι καλύτερο. Από εκεί και πέρα. Ή θα αλλάξετε το σημείο στο κείμενο που θα περιλάβετε αυτή την αναφορά ή θα με βρείτε αντίθετη. Τώρα, ε, στο 12, στο άρθρο 12, κάνετε λόγο για τις σελίδες, των, τις διαδικτυακές τοποθεσίες των αρμοδίων τμήματων της Επιτροπής. Αντί λοιπόν να βάλουμε την ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Αλίας, να βάλουμε τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ ή θα βάλουμε όλα τα τμήματα και υποτμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι λίγο υπερβολικό να αλλάξει το Γενική Διεύθυνση Αλληλείας και να γίνει ε, Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Υποθέσεων και το καθεξής. Μάρε δηλαδή. Γιατί όμως να βάλουμε την ξεχωριστή διαδικτυακή τοποθεσία ή στο σελίδα κάθε τμήματος και κάθε υποδιεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός και αν δεν κατάλαβα καλά τι γράφει το κείμενο. Τώρα, για όλο αυτό το θέμα του 75% συμφωνώ με τους συναδέλφους, άρα δεν θα κάνω περαιτέρω σχόλια. Και τελευταία παρατήρησή μου είναι η εξής. Στο άρθρο 22, στην ε, εισαγωγική διατύπωση, έχετε διαγράψει τον όρο «αλλιευτικά» από τα δεδομένα. Νομίζω ότι όταν μιλούμε για βασικά στοιχεία, βασικά δεδομένα, θα πρέπει να παραμείνει ο επιθετικός προσδιορισμός αλλιευτικά. Γιατί θέλετε να το διαγράψετε. Επί της αρχής δεν συμφωνώ με αυτή τη διαγραφή. Αυτές είναι οι γενικότερες παρατηρήσεις, τα γενικά σχόλια που θα ήθελα να κάνω. Να δώσω το λόγο στην Επιτροπή, στον κύριο Τζόνστον. Um, Ευχαριστώ. Και εμείς καλωσορίζουμε αυτή την έκθεση του εισηγητή και θεωρούμε ότι πολλές από τις τροπολογίες που προτείνονται είναι χρήσιμες. Πιστεύω ότι κινούμαστε προς τη κατεύθυνση σε ό,τι αφορά το να βρούμε ε, ένα κοινό παρανομαστή με το Συμβούλιο, το οποίο έχει συζητήσει, όπως ξέρετε, πολλές φορές αυτή την πρόταση και έχει υποβάλει κάποιες τροπολογίες. Ε, αυτές οι τροπολογίες κάπου συγκλίνουν με τις τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής. Διάφοροι ομιλητέ ε, εξέφρασαν ανησυχίε για την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότηση από 50% στο 75% και φυσικά αυτή η αύξηση συνδέει και τον έλεγχο, αφορά και τον έλεγχο και την εφαρμογή και την συλλογή των δεδομένων. Δεν θα σε εκπλήξει ότι και εμείς συμμεριζόμαστε αυτές τις ανησυχίες για τους λόγους που ακούστηκαν σήμερα εδώ. Αν δώσουμε ένα πολύ απλό παράδειγμα στον έλεγχο, για τον έλεγχο και την εφαρμογή. Έχουμε ας πούμε 100 ε, ευρώ συγχρηματοδότηση από τον κοινοτικό προπολογισμό και αυτό είναι το 75% του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι θα ξοδέψουμε 133 ευρώ συνολικά για προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται και από την κοινότητα και από τις εθνικές αρχές. Αν η συγχρηματοδότηση είναι 50% και έχουμε 100 ευρώ, θα ξοδέψουμε 200 ευρώ για αυτά τα προγράμματα. Επομένως, η αρχή μας είναι ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια αρχή χρηστής οικονομικής διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι σεβόμαστε τις αρχές οικονομίας. Αυτό τι σημαίνει, θα πρέπει να διαθέσουμε τους απαραίτητους ε, πόρους ε, έγκαιρα και τους πόρους που χρειαζόμαστε. Επομένως, θα έλεγα ε, να μην μειώσουμε το ποσοστό του ελέγχου, τα ποσά του ελέγχου αυξάνοντας το ποσοστό συγχρηματοδότησης. Το ίδιο και για τα υπόλοιπα στοιχεία. Τώρα, για την τροπολογία 2. Υπάρχουν δύο σημεία που θα ήθελα να θέσω για την τροπολογία 2. Πρώτον, υπάρχει εισαγωγή του by the proper national authorities ε, από τις κατάλληλες εθνικές αρχές. Δεν νομίζω ότι προσθέτουν τίποτα αυτές οι λέξεις, αυτό που είχαμε στο κείμενο. Γιατί ποτέ δεν υπήρχε θέμα. Πάντα οι δικαιούχοι είναι οι εθνικές αρχές και αυτή είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Νομίζουμε λοιπόν ότι δεν βοηθάει αυτή η αναφορά. Σε άλλα σημεία επίσης, ε, στην τροπολογία, ε, έχουμε εξάλλου διάφορα εδάφια στην τροπολογία αυτή. Στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο έχουμε την λέξη ανάπτυξη, development. Καταλαβαίνουμε γιατί βάζετε τη λέξη αυτή στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο, αλλά στο τρίτο εδάφιο μιλάτε για την αγορά, ανάπτυξη και εξυγχρονισμό των μέσων ελέγχου. Αυτό, μιλάμε, αυτό τι υπονοεί, σκάφη και αεροπλάνα. Δεν θέλουμε να πληρώσουμε την τεχνολογία ανάπτυξης αεροπλάνων ή σκαφών. Μιλάμε για τέτοιες επενδύσεις. Γι' αυτό σας παρακαλώ προσοχή με αυτή τη λέξη γιατί θα μας δημιουργήσει δυσκολία. Καλωσορίζουμε την έκθεση συνολικά, αλλά έχουμε πρόβλημα με την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης, όπως σας είπα. Ο κύριος Φερέιρα. Φερέιρα για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ. για τη συγχρηματοδότηση. Ο σημερινός κανονισμός λέει ότι σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, τα χρηματοδοτικά κοινοτικά μέτρα, το ποσοστό συγχρηματοδότησης δεν μπορεί να ξεπεράσει το 50% των δαπανών, των επιλέξιμων δαπανών. Εγώ προτείνω να πούμε ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει το 75%. Εγώ δεν λέω λοιπόν ότι η συγχρηματοδότηση θα πρέπει να πάει υποχρεωτικά στο 75% για όλα τα προγράμματα. Θέλω να αφήσουμε ανοιχτή αυτή τη δυνατότητα για κάποια προγράμματα. Η Κομισιόν, όπως είπε και προηγουμένως, θα κρατήσει τη διακριτική ευχαίρεια, ούτως ώστε να προωθήσει τη διαχείριση που θέλει, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ποσό που έχει στη διάθεσή της. Αντίθετα λοιπόν από αυτά που υπόθηκαν από διάφορους συναδέλφους, δεν νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει κατά ανάγκη σε μείωση του αριθμού των δράσεων που θα χρηματοδοτούνται. Απλώς ορίζουμε ένα νέο ανώτατο ποσό. Και αντίθετα από αυτό που λέγεται τώρα στο σημερινό κανονισμό, που λέει ότι η συγχρηματοδότηση δεν μπορεί να ξεπεράσει το 50%, τώρα θα λέμε στον καινούριο κανονισμό ότι η συγχρηματοδότηση δεν μπορεί να ξεπεράσει το 75%. Και όπως είπα προηγουμένως, δεν σημαίνει αυτό ότι όλες οι δράσεις πρέπει να φτάσουν σε ποσοστό 75%. Απλώς αφήνουμε μεγαλύτερη ευχέρεια στην Κομισιόν για να χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα όταν χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά τα συμπληρωματικά στοιχεία. Αυτό είναι ένα τρόπο για να ενθαρρύνουμε την παρουσίαση περισσότερων υποψηφιωτήτων, δηλαδή υποψηφίων δράσεων και η Κομισιόν θα κάνει τη διαλογή ανάλογα με το τι υπάρχει στη διάθεσή μας, τι, τι, τι προσφέρεται, ας πούμε, ανάλογα με την προσφορά. Και σε ορισμένε περιπτώσει δίνουμε τη δυνατότητα να φτάσουμε σε ποσοστό σε χρηματοδότηση αυτών των δράσεων ύψου 75%. Αν ζητάμε τώρα περισσότερα, περισσότερη εμπλοκή των κρατών μελών και νομίζω το ζητάμε γιατί σημαίνει περισσότερα δεδομένα αυτό, αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να το πληρώσουμε. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να έχουμε ποσοστά συγχρηματοδότησης υψηλότερα σε σχέση με τα σημερινά, σε σχέση με το 50%. Αυτό το λέω στην πρόεδρο σε σχέση με αυτά που είπε. Εσείς μιλούσατε για άρθρα, όχι για τροπολογίες, επομένως δεν ξέρω αν σας παρακολούθησα 100%, δεν ξέρω για ποια σημεία μιλούσατε. Αν κατάλαβα καλά, πάντως πρόεδρε, αυτά έχω να πω. Ε, τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ δεν τον, δεν τον έχουμε αντικαταστήσει. Τη Γενική Διεύθυνση Αλίας, δηλαδή. Γιατί δεν θέλουμε να συμβεί αυτό που συνέβη όταν ε, κάναμε την αλλαγή από το DG ε, Αλία σε DG Mare. Εδώ δεν εννοούμε την DG Mare. Πριν υπήρχε η DG Αλία. Τώρα είναι η DG Mare. Αύριο μπορεί να προκύψει κάτι άλλο. Αν κάνουμε αυτή την αναφορά, στην DG Mare δηλαδή, θα πρέπει να κάνουμε συνεχείς προσαρμογές των κειμένων. Μπορεί η Κομισιόν να αλλάξει το όνομα και μπορεί να προκύψει κάτι άλλο. Επομένω, ο κανονισμό δεν θα είναι επίκαιρο αν με το μετονομαστεί Mare. Γιατί θα αναφέρεται σε κάτι που δεν θα υπάρχει πια. Επίσης, διαγράψαμε το δεδομένα αλίας. Εδώ μιλάμε για δεδομένα. εμεί θέλουμε μάλλον να μιλήσουμε και για δεδομένα αλλία και για δεδομένα καλλιέργεια. Μια και μιλάμε ούτως ή άλλως για την υδατοκαλλιέργεια. θέλαμε να συμπεριλάβουμε και την υδατοκαλλιέργεια. Αυτά σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Τζόνστον. Θέλω να σας πω το εξής. Οπου, οποτεδήποτε μιλάμε για αγορά των κρατών μελών οποιοδήποτε εξοπλισμού, Πάντοτε μιλάμε για αγορά μιλάμε και για ανάπτυξη. Ε, ανάπτυξη τεχνολογία, ανάπτυξη εξοπλισμού κτλ. Δεν θέλουμε μόνο να, αγοράζει, αγοράσουν τα κράτη-μέλη, θέλουμε να, προωθήσουν, θέλουμε να προωθήσουν και την τεχνολογία. Γιατί λοιπόν να μην χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας, αν υπάρχει περι, περιθώριο ανάπτυξης. Γιατί να χρηματοδοτούμε μόνο την αγορά και όχι την ανάπτυξη της τεχνολογίας, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή η τεχνολογία. Το κάνουμε και σε άλλους τομεί. γιατί όχι εδώ. Η αγορά και ο εξυγχρονισμό των μέσων ελέγχου. Ωραία, χρηματοδοτούμε την αγορά. Γιατί να μην χρηματοδοτήσουμε και την ανάπτυξη αυτού του, των μέσων, αυτού του εξοπλισμού υποχρέωση που βαραίνει τα κράτη-μέλη. Αυτά. Νομίζω ότι απάντησα και αν κάτι ξέχασα είμαι στη διάθεσή σα. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξαναπάρει το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Τζόνσον. Ναι, να σχολιάσω αυτό το τελευταίο σημείο για τις αγορές των σκαφών και των αεροσκαφών. Δεν είμαστε αντίθετοι με την ιδέα ότι για, το υπό, για τους υπόλοιπους ελέγχους θα πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη. Προφανώς θα πρέπει να το δούμε αυτό, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό, αλλά αν μιλήσουμε για τις, για τις αγορές σκαφών για περιπολίες και των αεροσκαφών, ε, θα πρέπει όντως να έχουμε περισσότερα, να δώσουμε περισσότερα, γιατί εσείς μιλάτε για χρήματα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα για το πρόγραμμα αυτό. Μιλούμε για πρόγραμμα που έχει κορδίλει 45 εκατομμύρια το χρόνο σύμφωνα με τη δημοσιονομική προοπτική. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το αντέξει αυτό το πρόγραμμα. Η ανάπτυξη των ελεγκτικών μηχανισμών και τεχνολογιών, η ανάπτυξη, η αγορά των ε, σκαφών και αεροσκαφών για περιπολίες θα πρέπει να γίνει μέσω των επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε αυτό το τομέα. Και αν πρέπει να υπάρξει επιστημονική ανάπτυξη, θα πρέπει να γίνει μέσω ενό επιστημονικού προγράμματος. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτό μπορεί να γίνει σε τούτο εδώ το πρόγραμμα. Και ε, για την αύξηση από το 50% στο 75%. Είναι σαφές ότι αυτό που λέει ο συγκητής είναι ότι δεν υποχρεούμεθα να δώσουμε 75% σύμφωνα με την ε, έκθεση. Αυτό ισχύει. Αλλά δεν πρέπει να υποτιμούμε και τις ε, προσδοκίες που θα δημιουργηθούν στα κράτη-μέλη εάν θέσουμε ένα ε, ποσοστό 75% σε έναν κανονισμό. Ε, Πολλέ φορέ έχουμε ξεπεράσει τις, ε, το 50% ας πούμε για τι νέε τεχνολογίε. Και όταν τέθησε ισχύ ο νέο κανονισμό για τον έλεγχο υπήρξε δαπάνη κατά προτεραιότητα εκεί. Οπότε έχουμε ξεπεράσει ήδη και από πέρσι και φέτο το 50%. Και αυτό είναι ένα μηχανισμό ο οποίο θα παραμείνει και θα τον χρησιμοποιούμε, αλλά θέλουμε η αρχή, η έναρξη να γίνεται στο 50%. Καλώ. Ο κύριο Φερέιρα ε, για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Έχετε το λόγο. Ε, ε, Ένα πράγμα να υπογραμμίσω, κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, που αναγνωρίζει η Κομισιόν. Γιατί το ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι. Αν αυξήσουμε το ποσοστό από το 50% στο 70%, αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνεται ο αριθμός των δράσεων που χρηματοδοτούνται. Αυτό να το ξεκαθαρίσω. Φυσικά, με αυτόν τον τρόπο ε, μπορεί να δημιουργηθούν διάφορες προσδοκίες, αλλά θα δημιουργηθούν και περιθώ... μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι καλό για την συλλογή και διάδοση δεδομένων. Αγαπητέ συνάδελφε Φερέιρα, σε δύο παρεμβάσεις ακούσαμε ότι η Κομισιόν δεν ενδιαφέρεται καθόλου να αυξήσει το ποσοστό συγχρηματοδότησης. Οπότε γιατί πρέπει να, τους, ε, να, να σας κάνουμε αναγκαστικά τη χάρη. Η Κομισιόν λέει όχι. Ε, Νομίζω ότι έχει επιχειρηματολογήσει πολύ καλά και έχει δικαιολογήσει πολύ ε, σωστά ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ότι δεν είναι προς όφελος όλων η, αύξηση της χρηματοδότησης. Εδώ γίνονται κάποιες ε, κάποια αιτήματα και ε, το θέμα είναι πάντα πώς θα διατυπώνουμε αυτά τα αιτήματα. Ε, σε εγώ προέρχομαι από μια χώρα όπου τέτοια, αυτά τα αιτήματα δεν ε, χρειάζονται και πολλές πολλές φιωριτούρες για να γίνουν πραγματικότητα. Αν τώρα ε, θέλετε να αυξηθεί η χρηματοδότηση στο 75% ε, θεωρώ ότι στο τέλος όλα τα αιτήματα θα διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνουν ε, συγχρονοδότηση 75%. Δεν νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση στο μέλλον να μπορέσουμε να χρηματοδοτούμε τον έλεγχο στο 75% που ζητάτε εσείς. Και εκεί το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Σας ζητώ λοιπόν να το ξανασκεφτείτε. Για τις πλούσιες χώρες ε, αυτό θα είναι μικρό, μικρό πρόβλημα. Αλλά αν σε έναν ε, κανονισμό μπει γραπτό το 75% ότι θα υπάρξει τόση πολλή φαντασία στα αιτήματα των υπολείπων χωρών που όλοι θα θέλουν 75% χρηματοδότηση. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι οι δύο θέσεις είναι σαφέστατες. Ο κύριος Φερέιρα έχει εκθέσει επαρκώς τη δική του, η Επιτροπή έχει εκθέσει επαρκώς τη δική της. Εσείς έχετε τον τελευταίο λόγο, κύριε Φερέιρα, ως εισηγητής, αν θέλετε να πείτε κάποιο καταληκτικό σχόλιο. Σύντομα, Πρόεδρε. Δεν θέλω να υπάρχουν παρεξηγήσεις και αμφιβολίες. Η, η συνάδελφος είπε ότι ήρθε εδώ η Επιτροπή για να υπρασπιστεί μία θέση. Όντως. Πάντως ακούσαμε διάφορα από διάφορους συναδέλφους διάφορα επιχειρήματα αλλά δεν θέλω όμως ε, να πάρετε τη λάθος απόφαση βασιζόμενη σε λάθος στοιχεία. Αυτό είναι το θέμα, γιατί συχνά το σημείο εκείνης σας ήταν λάθος. Έχουμε πει κατ' επανάληψη τη σημασία απόκτησης επιστημονικών δεδομένων και έχουμε επίσης πολλές φορές μιλήσει για τη σημασία του ελέγχου. Επίσης έχουμε αγωνιστεί για να έχουμε τους απαραίτητους πόρους για τον τομέα της αλίας εν γέννη και για τους δύο υποτομείς που σας ανέφερα. Στα πλαίσια της συζήτηση που κάνουμε για τον προϋπολογισμό και για τις δημοσιονομικές προοπτικές, καλό θα ήταν η Επιτροπή μας να στείλει ένα μήνυμα και να πει ότι υπάρχουν τομείς που πρέπει να τους προσέξουμε ιδιαίτερως. Νομίζω ότι αν κάνουμε αυτό που λέω θα δώσουμε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα ως Επιτροπή. Μπορεί τελικά να οδηγήσει σε αύξηση ή όχι των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας σε αυτόν τον τομέα. Η Κομισιόν μπορεί να κάνει την διαχείριση που επιθυμεί και με τους ίδιους πόρους. μπορεί να συνεχίσει τη διαχείριση που ασκεί σήμερα, ας πούμε. Απλώς θα είναι ξεκάθαρα όλα αυτά. Καλώς. Όλοι λοιπόν έχουν διαμορφώσει πλέον την άποψή τους. 9 Νοεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών και θα ψηφίσουμε ή στις 30 Νοεμβρίου ή την 1η Δεκεμβρίου σε αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ολοκληρώνεται λοιπόν η εξέταση του σημείου 9 της ημερήσιας διάταξης και περνούμε στο 10 συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χιλής για τη διατήρηση των αποθεμάτων του Ξηφία στο νοτιοανατολικό ειρηνικό ωκεανό. Η συγητής είναι ο κύριος Γκάλαχερ. Εγώ δεν ήμουν παρούσα στην τελευταία συνεδρίαση, προέδρευσε ο κύριος Στίβενσον. Η σοσιαλιστική ομάδα ζήτησε να το ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό, επομένως γι' αυτό και δίνω το λόγο στον εισηγητή και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Δεν μπόρεσα να παραστώ στην τελευταία συνεδρίαση, αλλά η επεξηγηματική μου δήλωση ε, παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση που, όπου έλειπα. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Κομισιόν με προσκάλεσε να συμμετάσχω σε μία διάσκεψη. Το έκανα. Και μου δόθηκαν διάφορες εξηγήσεις δεν θέλω να επανέλθουμε σε παλιές ιστορίες. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ελήφθησαν αποφάσεις πριν από την πρώτη συνεισφορά της Κομισιόν για το θέμα αυτό. Ε, κάποια στοιχεία ήταν διαθέσιμα ε, σε μια άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά όχι σε εμά. Τέλο πάντων, α τα αφήσουμε αυτά κατά μέρο. Πιστεύω, πιστεύω όμω ότι κανονικά μία υπεύθυνη κοινοβουλευτική επιτροπή θα έπρεπε να μας ενημερώσει. Όχι, δεν υπάρχει νομική υποχρέωση, άλλου τύπου υποχρέωση. Είναι παλιός ο φάκελος αυτός, πάνω από 10 χρόνια. Ε, διαπιστώσαμε εδώ και 10 χρόνια ότι δεν συνεργάζονταν οι χιλιανοί, ε, ότι είχαν μονομερή στάση για τα αλλιεύματα, στα νερά τους, για τις εκφορτώσεις, ε, στα λιμάνια της Χιλής για λόγους που εκείνοι καταλαβαίνουν. Εγώ δεν καταλαβαίνω πάντως. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα ευρωπαϊκά σκάφη δεν μπορούσαν να μπουν στη Χιλή. Έπρεπε να πάνε στο Περού δηλαδή ή να μεταφορτώσουν μέσα σε επικίνδυνες συνθήκες. Στην ανοιχτή θάλασσα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό αρχικά υπήρχε μια ενδιάμεση συμφωνία. Αλλά ακόμα εκεί η ενδιάμεση συμφωνία δεν λειτουργήσε ποτέ. Δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης. Ποτέ. Και ούτω ή άλλω κάλυψε μόνο τέσσερα σκάφη τα οποία θα μπορούσαν να είχαν πρόσβαση στην Χιλή. Δεν έχει νόημα. Δεν είχε νόημα αυτή η ενδιάμεση συμφωνία. Πριν από το καλοκαίρι, εγώ δεν είμαι πεπισμένο ότι σκόπευε να συνεργαστεί η Χιλή. Ε, για το, και για το θέμα του ξεφία. για να το πω ομά, πιστεύω ότι η χιλή απλώς καθυστερεί από χρόνο σε χρόνο. Εγώ και στα περιφερειακά συμβούλια ε, και ο κύριος Στίβενσον συναντήθηκα με τους αξιωματούχους του Περιφερειακού Συμβουλίου στο, Άστερ, στο Άμστερνταμ και τα λοιπά και ενημερώθηκα ότι δεν αφορούσε μόνο το θέμα αυτό το ξηφία αλλά και άλλα αποθέματα όπως το σαφρίδι και άλλα θέματα και άλλα δηλαδή αποθέματα. Υπάρχει πρόβλημα. Οι αρχές της Χιλής είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν και μονομερός και διμερός με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλες χώρες που δραστηριοποιούνται στον νότιο ανατολικό ειρηνικό. Εμείς πρέπει να πάρουμε την απόφαση ως Επιτροπή και συνεχεία το Κοινοβούλιο συνολικά. Αν αποφασίσουμε να μην εγκρίνουμε το σημείο αυτό, τότε η Κομισιόν θα πρέπει να μας παρουσιάσει εναλλακτικέ ε, προτάσεις. Στο παρελθόν, όταν δεν υπήρχε συμφωνία, μπορούσαμε να προσφύγουμε στον ΠΟΕ. Την τελευταία φορά, όταν το θέμα ε, έφτασε στην Επιτροπή, αυτή την άποψη είχα. Πριν από χρόνια. Δεν έχω πιστικά επιχειρήματα που με πείθουν ότι ήγηκε η ώρα να αλλάξω τις συστάσεις μου προς την Επιτροπή. Δηλαδή, μου είπαν ότι η στάση κάποιων αλλιέων στην Ισπανία έχει αλλάξει, αλλά δεν βλέπω τίποτα που να με πείθει ότι θα πρέπει εγώ να σας συστήσω να να αλλάξετε στάση. Δηλαδή ότι θα πρέπει εγώ, εν πάση περιπτώσει, να αλλάξω την σύστασή Εγώ συστάσει κάνω. Αυτό που αποφασίζει είναι η Επιτροπή. Σω υπάρχουν και άλλα μέλη τη Επιτροπή, άλλοι βουλευτέ που να γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση. Εγώ όμω τα έχω μελετήσει τα πράγματα. Συζήτησα με την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Εννοώ Επιτροπή και συζήτησα και με, τους, με άλλου. Ε, στο παρελθόν υπήρχε λογική μην κάνει τίποτα αν δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί, να ανοίξουν, εν πάση περιπτώσει, τα λιμάνια της Χιλής μόνιμα. Όχι να βρούμε μία προσωρινή λύση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Η κυρία Αντρές Βάρεα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχει δίκιο σε αυτά που λέει ο κύριος Γκάλαχερ. Όντως ασχολούμαστε με το θέμα αυτό τα τελευταία δέκα χρόνια τουλάχιστον και πρόκειται για εμπορικό εμπόδιο στις ε, μεταφορτώσεις και εκφορτώσεις σε σχέση και με τη χιλή. Η μονομερής εφαρμογή ε, των δικών της ε, κανόνων της χιλής είναι ένα από τα προβλήματα και όντως υπήρξε αντιπροβλήματα. Ωστόσο, μία τέτοια συμφωνία ουσιαστικά βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χιλής, ακόμα και αναφορά σε ένα μόνο ψάρι, τον ξηφία εφαρμόζονται διεθνείς πρακτικές και η Χιλή μέχρι σήμερα δεν ε, εφήρμοζε κανένα είδος ε, κανόνα και κανονισμού και τώρα πλέον έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει ε, τέτοιου είδους διεθνείς πρακτικές. Τώρα, για τις μεταφορτώσεις. Όπως το είπε και το κύριος Γκάλαχερ, και εγώ πιστεύω ότι έχει λυθεί το θέμα. Αυτό πιστεύει και ο κλάδος άλλωστε και μπορούν να γίνουν μεταφορτώσεις και εκφορτώσεις χωρίς προβλήματα. Δεν πρέπει να μείνουμε όμως αυτό θα πρέπει η Χιλή να προσχωρήσει σε μια διεθνή κανονιστική νομοθεσία για τη δεντολογία, για τον τρόπο συμπεριφοράς αν θέλετε, για τη διαχείριση, για την τήρηση και εφαρμογή τέτοιου είδους κριτηρίων και προϋποθέσεων. Εάν δεν υπογράψουμε μια τέτοια συνθήκη, μια τέτοια συμφωνία, τότε ποτέ η Χιλή δεν πρόκειται να εφαρμόσει θέντα και άρα ποτέ δεν θα αποτελέσει μέλος των πολυμερών διαβουλεύσεων για τα υφιστάμενα αποθέματα. Δεν εντάσσεται σε κανένα περιφερειακό γνωμοδοτικό συμβούλιο η χώρα αυτή και δεν ανήκει και στο Διεθνή Οργανισμό για την Αλία. Επομένως, έχοντας σημαντική παράκτια ζώνη, όντας μια σημαντική χώρα ενδυνάμει για την Ευρώπη, όντας ένα σημείο γέφυρας θα έλεγα, καλό θα ήταν να υπογράψουμε μια συμφωνία με τη χώρα αυτή. Είναι μια πρόοδος είναι κάτι που θα ωφελήσει και τα δύο μέρη. Δεν μπορεί κανείς να μένει στο περιθώριο. Όντως η Χιλή δεν έχει εφαρμόσει αυτά που θα έπρεπε. Ωστόσο, ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και αυτός. Δηλαδή, χώρες που δεν μπαίνουν ε, στην ε, διεθνή συνύπαρξη αν θέλετε, τουλάχιστον να εκπληρώσουν κάποιους ε, κανόνες, κάποιες προϋποθέσεις. Κάποιες προϋποθέσεις. Τώρα, εάν υπογράψουμε και τελικά η Χιλή δεν τηρήσει τα δέοντα και τα ε, πεπραγμένα, έχουμε τρόπους να ε, σημάνουμε αυτό το καμπανάκι. Ή αλλιώς θέτουμε σε χειρότερη μοίρα τον Ισπανικό αλλιευτικό στόλο και εν συνολικά τον Ευρωπαϊκό αλλιευτικό στόλο. Σίγουρα θα ακούσουμε και απόψεις αντίθετες. Εγώ όμως μιλώ για έναν τρόπο επίτευξης μιας διεθνούς συμφωνίας, η οποία ακριβώς θα έχει αυτό το σκοπό, να δεσμεύει και τα δύο μέρη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο κύριος Γκιάγκικ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω εξ αρχής ότι Συμφωνώ απολύτως και στηρίζω τον εισηγητή, ο οποίος εξ ονόματο της Επιτροπής Αλίας αποφάσισε να απορρίψει την ε, ε, συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Χιλής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σχέδια μη πρόσβαση στους λιμένες αποσύρθηκαν και δεν έχουμε βελτίωση ε, στους χιλιανούς λιμένες, στην κατάσταση εκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι με τη συμφωνία του 2008 όλος ο ευρωπαϊκός στόλος έχει τη δυνατότητα να εκφορτώσει στους χιλιανούς λιμένες χωρίς παρατηρητές, ωστόσο η Χιλή δεν έχει εφαρμόσει τα πρότυπα τα ευρωπαϊκά και λαμβάνονται μέτρα διατήρησης για πρώτη φορά για τον ξηφία στο νότιο ανατολικό ειρηνικό. Όμως δεν έχω δει κανένα κείμενο που να εγγυάται κάτι τέτοιο. Δεν πιστεύω ότι θα τηρήσει η χιλή της δεσμεύσης της γιατί δεν το έχει κάνει ποτέ μέχρι σήμερα. Δεν είναι μόνο συμβολικός αυτός ο, ε, συμβολική αυτή η απόρριψη ε, της συμφωνίας νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ε, προς τη χώρα αυτή. Η κυρία Λέβιν, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο ε, για τη γενικότερη διαμάχη για το θέμα του, του ξηφία. Οι χιλιανοί λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σέβεται τα ελάχιστα μεγέθη για τις εκφορτώσεις που εφαρμόζουν αυτοί και ότι εμείς έχουμε άλλα μεγέθη και ότι αυτό είναι το σημείο από όπου ξεκίνησε και η διαμάχη. Θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω αυτό το γενικότερο πρόβλημα της απουσίας συντονισμού από τη δική μας πλευρά στο διεθνές στερέωμα ώστε να λύνονται τέτοιου ζητήματα στους κόλπους των περιφερειακών οργανώσεων αγοράς και των περιφερειακών συμβουλίων. Όντως η χιλή δεν είναι ε, μέρος του αρεθμό για τον τροπικό τόνο και αυτό είναι, αυτό είναι και η βάση αν θέλετε του προβλήματος δηλαδή η αλίευση του ξηφία εκτός χιλής είναι πρόβλημα γιατί η αλίευση του, ξηφία είναι ε, άναρχη και αρρύθμιστη. Δεν είναι λαθρέα αλληλεία απαραίτητα, αλλά είναι σίγουρα άναρχη, δεν υπόκειται σε κανονιστικές διατάξεις. Και αυτό ε, θα πρέπει να το υπογραμμίσω και ελπίζω στην επικείμενη έκθεσή μου για την παράνομη, άναρχη και λαθρέα αλία να είμαι σε θέση να το ε, τονίσω ακόμα περισσότερο και να το αναδείξω το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, δεν ξέρω να μιλήσω ή να σοπάσω. Βεβαίως στηρίζω τον εισηγητή. Ωστόσο, καλύτερα να σοπάσω, γνωρίζετε τη θέση μου, να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ε, άλλωστε ένα θέμα που προκύπτει από την καλή θέληση της χιλής. Ο πελαγικός στόλος αντιμετωπίζει τις ίδιες συνθήκες με το στόλο που αλλιεύει τον Ξηφία. Εγώ έχω μιλήσει με τον διευθυντή που είναι Ολλανδός, δεν είναι Ισπανός και Ήθελα να το επιβεβαιώσω και το επιβεβαίωσα δηλαδή ότι ακόμα και για αλλαγή πληρώματος πρέπει να κάνουν ταξίδι 8 ημερών μέχρι να φτάσουν ε, στο χείλη του Περού για να αλλάξουν πλήρωμα. Και με αυτή την έννοια ο πελαγικός στόλος αλλιεύει πέρα από τα ύδατα που εντάσσονται στην αρμοδιότητα της χιλής, αλλιεύει στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά και ο στόλος που αλλιεύει τον ξηφία αλλιεύει στην ανοιχτή θάλασσα, πέρα από τα ύδατα αρμοδιότητας της χιλής και ωστόσο ούτε για να αλλάξουν πλήρωμα δεν τους επιτρέπουν οι χιλιανοί να σταθμεύσουν στους λιμένες με αυτο, τους χιλιανούς με αυτό το σκοπό. Λοιπόν, η κυβέρνηση της Χιλής έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα και δεν έχει υπάρξει καμία παρέκκληση από τα διατάγματα που έχει εκδώσει η κυβέρνηση της Χιλής. Επομένως, εάν πρόκειται για θέμα συμμόρφωσης ε, με το διεθνές δίκαιο, τότε μπορούμε να απαιτήσουμε αυτού του είδους τη συμμόρφωση. Δεν χρειαζόμαστε μνημόνιο. Και μάλιστα το αναστήλαμε στο παρελθόν διότι η χιλιανή πλευρά δεν τηρούσε ε, το διεθνές δίκαιο. Είναι θέμα καλής θέλησης απλά, να έχουν τη βούληση. Και εκφράζω αυτό το παράπονο ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας έχουν κοροϊδέψει. Εμάς εδώ στην Επιτροπή Αλίας. Ενδεχομένω όχι στην Επιτροπή για το Διεθνέ Εμπόριο, αλλά σίγουρα ναι εδώ στην Επιτροπή Αλληλεία. Το 2002 θα θυμάστε ότι αναστάλθηκε η προσφυγή που είχε κατατεθεί ενώπιον του ΠΟΕ με πρόφαση το περιβόητο μνημόνιο, το οποίο τελικά δεν εγκρίθηκε, δεν υπογράφτηκε και δεν επικυρώθηκε ποτέ. Και η αρμόδια επιτροπή το απόσυρε εκ των προτέρων πριν προχωρήσουμε στην κύρωση αυτής της συμφωνίας. Άρα ήταν κοροϊδία. Μας κοροϊδέψαν. Δεν θα είχαμε αποσύρει την προσφυγή μας στον ΠΟΕ. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ απολύτω με τον εισηγητή. Δεν νομίζω ότι οι χιλιανοί έχουν σκοπό να κάνουν κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι το θέμα ε, του αλληλευτικού στόλου για τον Ξηφία. Είναι για το σύνολο του αλληλευτικού στόλου που δραστηριοποιείται στην ανοιχτή θάλασσα. Επομένως, εγώ συμφωνώ πλήρως, στηρίζω απολύτως, με τον, στηρίζω απολύτως τον εισηγητή. Θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να εκφράσουμε ξεκάθαρα την αντίρρησή μας. Και δεν νομίζω ότι ούτε θα βελτιωθούν, ούτε θα επιδεινωθούν με την άρνησή μας αυτή οι διεθνείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Χιλή, οι οποίες κατά τα λοιπά είναι πολύ καλές. Ο κύριος ε, Γκρίμο μας ακούει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους διάφορους ομιλητές που πήραν το λόγο για αυτή την ενδελεχή συζήτηση που κάνουμε για το θέμα αυτό. Όπως σημειώθηκε από τον εισηγητή, τον κύριο Γκάλαγκερ, το θέμα είναι περίπλοκο. Και ελπίζω ότι το ενημερωτικό σημείωμα το οποίο διενεμήθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα μέλη της ε, κοινοβουλευτική επιτροπή σα θα είναι χρήσιμο για να βελτιώσετε την κατανόηση του θέματος. Τουλάχιστον την κατανόηση αυτών που δεν γνωρίζουν το θέμα τα τελευταία δέκα χρόνια. Αυτό είναι λοιπόν το περίπλοκο πλαίσιο. Ε, υπάρχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες. Υπάρχουν τα οικονομικά ευρωπαϊκά συμφέροντα, υπάρχουν τα θέματα τη διατήρηση των αποθεμάτων και υπάρχει και το θέμα των σχέσεών μας με τη Χιλή. Κατά την άποψη τη Κομισιόν, οποιαδήποτε και είναι η οπτική γωνία, το συμπέρασμα είναι το ίδιο. Αν κοιτάξουμε τα οικονομικά ευρωπαϊκά συμφέροντα καταρχήν σε σχέση με την διευθέτηση του 2001, δεν υπάρχουν ε, πλέον περιορισμοί για τις, πορτο, για τις ποσότητες ε, που εκφορτώνονται, δεν υπάρχουν όρια για τα σκάφη, δεν υπάρχει μονομερής εφαρμογή ε, κανένας μέτρου από τη Χιλή ε, της νομοθεσίας της για το ελάχιστο μέγεθος του ξηφία είναι αυτό το μνημόνιο, αυτό το understanding ε, φέρνει σημαντικές ε, βελτιώσεις σχέση με τα όσα είχαμε συμφωνήσει το 2001. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα, η συμφωνία είναι ενδιαφέρουσα. Γι' αυτό ακριβώς ο τομέας ε, είναι υπέρ της, υποστήρι... είναι υπέρ της ε, συμφωνίας αυτής. Τώρα, για τη διατήρηση των πόρων. Κάτι που μας ανησυχούσε επίσης. Αυτή η συμφωνία έχει διατάξεις για να εφαρμόσουμε ένα πάγωμα για τον αριθμό των σκαφών που ψαρεύουν ε, ξηφία. Είναι ένα από τα πρώτα μέτρα ε, διατήρησης του ξηφία στο νοτιοανατολικό ειρηνικό. Είναι ένα μέτρο ακόμα για να βοηθήσουμε την καλύτερη διατήρηση του είδους αυτού. Δεν ξέρω αν είναι επαρκή, δεν ξέρω αν χρειάζεται και άλλα μέτρα. Αλλά αν δεν επικυρώσουμε αυτή τη ε, συμφωνία σήμερα, δεν θα έχουμε τίποτα στα χέρια μα. Αν επικυρώσουμε, θα έχουμε ένα μέτρο διατήρηση, αλλά αν δεν την ε, επικυρώσουμε, θα έχουμε τίποτα για τη διατήρηση του ψηφία. Η αρμόδια περιφερειακή οργάνωση Ελία για τη διαχείριση και διατήρηση και διαχείριση του ψηφία και των τονοειδών έχει, έχει το εξή πρόβλημα, ότι η Χιλή δεν είναι μέλος της. Και τώρα πάω στο τρίτο θέμα. Η Χιλή τα τελευταία χρόνια έχει δείξει μια προθυμία, για να μην πω κάτι περισσότερο, για να δεσμευτεί στη, στα πλαίσια μιας διεθνούς συνεργασίας με σκοπό την πρόθεση της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων. Μέσω της ε, διαπραγμάτευσης νομίζω ότι μπορούμε να εξαναγκάσουμε τη Χιλή να εμπλακεί περισσότερο ε, σε διεθνές πλαίσιο. Μέσω της διμερούς αυτής συμφωνίας ή κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός. Ε, και νομίζω ότι τη βοηθάμε να δεχτεί, ε, να κάνει κάποια ανοίγματα για την πρόσβαση στα λιμάνια της. Επίσης, για πρώτη φορά η Χιλή συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις που έγιναν για να θεσπίσουμε μια νέα οργάνωση στον νοτιοανατολικό ειρηνικό. Γιατί παλιά δεν υπάρχει πια. Δείχνει λοιπόν ότι αλλάζει ε, Στάση Χιλή παλιά δεν ήθελε να συμμετάσχει σε αυτή την οργάνωση, τώρα όμω κάνει κάποια βήματα προ αυτή την κατεύθυνση. μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν αρκεί αυτή η προσπάθεια. Το, ε, το θέμα πάντως είναι ότι όταν η Χιλή κάνει βήματα μπορούμε, θέλουμε να, τα, να την εθαρρύνουμε. Γιατί μέσω αυτής της διμερούς συμφωνία θα έχουμε μια διμερή Επιτροπή για να κοιτάμε κατά πόσο εφαρμόζεται η συμφωνία και θα έχουμε ένα μηχανισμό επίλυσης, διμερή μηχανισμό επίλυσης ε, διαφορών, αν θεωρήσουμε ότι η Χιλή δεν συμμορφώνεται. Επίσης μπορούμε να την πιέσουμε για να ασχοληθεί περισσότερο με την ε, βιώσιμη διατήρηση. Αυτή είναι η επιλογή. Αν ε, απορρίψετε αυτό που προέκυψε από τη διαπραγμάτευση, δεν ξέρω ποιε είναι οι εναλλακτικέ λύσει. Υπάρχουν ιδέες Φυσικά αν υπάρχουν, η Κομισιόν θα ήθελε να τι ακούσει αυτές τις ιδέες, αλλά σε αυτή τη φάση η Κομισιόν δεν γνωρίζει σε ποιο βαθμό η απόρριψη της συμφωνίας μπορεί να οδηγήσει στην βελτίωση της ε, κατάστασης των Ευρωπαίων αλλιέων, που νομίζω ότι θα είναι τα πρώτα θύματα από την απόρριψη της συμφωνίας. Δεύτερον, δεν ξέρω αν απορρίψουμε τη συμφωνία, αν θα βελτιώσουμε την διατήρηση των αποθεμάτων. Σκεφτείτε το. Τρίτον, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό η απόρριψη αυτής της συμφωνίας θα επέτρεπε ε, στη Χιλή να κάνει περισσότερα βήματα για τη διμερή συνεργασία και να την αναγκάσει να γίνει πιο αξιόπιστος εταίρος, ε, πιο συνεργάσιμος εταίρος από ό,τι στο παρελθόν. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως, ε, μου άρεσε το γεγονός ότι βάλατε αυτό το θέμα στην διατάξη. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και για τα ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα, αλλά και για την προσπάθεια που κάνουμε εμείς για την ε, διατήρηση και διαχείριση των αποθεμάτων στο νοτιοανατολικό ειρηνικό κενό. Ευχαριστώ. Αν δεν θέλει να προσθέσει κάτι ο κύριος Γκάλαχερ, να κλείσουμε το θέμα αυτό. Να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τις απόψεις της και μόλις πάρουμε την ε, γνωμοδότηση θα μπορέσουμε έτσι να ωφελήσουμε την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και τις οικονομικές μας σχέσεις αλλά και γενικώ τις σχέσεις μας με τη Χιλή. Βεβαίω θα υπάρχει μια ομάδα που θα συνεργάζεται στενά με τη Χιλή για την ε, διατήρηση και θα υπάρξει και η διμερής ε, συμφωνία. Θα πιέσουμε λοιπόν την ε, Χιλή να ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό διατήρησης και αν αποφασίσουμε να μην δώσουμε την έγκριση, η Κομισιόν θα πρέπει να επανέλθει εδώ σε εμά και να μα δώσει μια εναλλακτική πρόταση εγώ θα πρότεινα να αποταθούμε στον ΠΟΕ και να περιμένουμε λίγο περισσότερο, μεν, αλλά ίσως αυτό να είναι ένα καλό μάθημα που τελικά έπρεπε να, να πάρουμε. Να μην κλείνουμε τη μία, τη μία πόρτα πριν, πριν ανοίξει η άλλη. Και αυτή τη στιγμή αυτό έχουμε κάνει. Οπότε ίσω θα έπρεπε να ε, εξασφαλίσουμε από την Κομισιόν, είτε τώρα είτε σε μια μεταγενέστερη φάση, ότι αν τελικά ε, στραφούμε στον ΠΟΕ, να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό και να δούμε και ποια είναι τα μειονεκτήματα των ε, ισπανικών σκαφών και των φορτώσεων που γίνονται σε μεγαλύτερα σκάφη και τα οποία μετά μεταφορτώνονται σε άλλα μεγαλύτερα σκάφη στον Ατλαντικό. Μιλούμε για κάτι πολύ απλό, υγεία και ασφάλεια. Μιλούμε για 68 μέρες στην ανοιχτή θάλασσα. Αν αυτό δεν σημαίνει συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, τότε εξηγήστε μου τι σημαίνει γιατί δεν καταλαβαίνω. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί εγώ πρέπει να αλλάξω την άποψή μας προς αυτό. Συμφωνώ απολύτως μαζί, απολύτως μαζί σας και τα λέτε και πολύ καλά. Τέλος πάντων, να κλείσουμε αυτό το θέμα. 9 Νοεμβρίου το μεσημέρι είναι η καταλεκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Άρα, ε, τροπολογίες διαδικαστικές θα γίνουν αποδεκτές μόνο. Επομένως, γνωρίζετε τη διαδικασία. οι τροπολογίες που θα γίνουν δεκτές ε, θα είναι μόνο διαδικαστικές, όπως γνωρίζετε. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την εξέταση του σημείου 10 της ημερήσιας διάταξης. Περνάμε στο 11, τροποποίηση του κανονισμού 1288 κάθετος 2009, σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών τεχνικών μέτρων από 1η Πρώτου του 10 έως 30 Ιουνίου του 11. Η κυρία Γκρελιέ είναι η συγγήτρια αυτό σχετίζεται άμεσα με τα τεχνικά μέτρα, με τον κανονισμό 850 και με την απόσυρση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Ιδία. Επομένως, 30 Ιουνίου του 2011 προτείνεται η παράταση, αν δεν απατώμε, να δώσω το λόγο στην κυρία Γκρελιέ να μας ενημερώσει και, μερά, και μετά εκπρόσωπο της Επιτροπής. Έχετε το λόγο, κυρία Κρελιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το 2008, όπως είπατε, η Κομισιόν έκανε μια πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τη συντήρηση των ληφτικών πόρων. Ε, Όμω η Κομισιόν και το Συμβούλιο δεν συμφώνησαν για τον κανονισμό αυτό για διάφορου λόγου και η πρόταση αυτή δεν υιοθετήθηκε. Η Κομισιόν, επομένως, προτείνει να ξαναδούμε τον κανονισμό σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο, στα πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτική πολιτική. Καταλαβαίνουμε αυτή την γενικότερη, σφαιρικότερη θεώρηση. Είναι ένα θέμα όμω που το δουλεύουμε από το 2008. Θα ήθελα λοιπόν η Κομισιόν να μα πει ποιε είναι οι προθέσει τη σε αυτόν τον τομέα. Γιατί ασχολούμαστε εδώ και παραπάνω από δύο χρόνια με αυτό το θέμα. Καταλαβαίνουμε βέβαια εσεί γιατί θέλετε να το εντάξετε σε ένα γενικότερο πλαίσιο, αλλά έχουμε και πολύ συγκεκριμένα σχόλια ενδεχομένω να κάνουμε λόγω του ότι είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με το θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια που ζητάει από την Κομισιό να εξηγήσουμε για ποιο λόγο παρατείνουμε αυτό το μηχανισμό στο πλαίσιο μιας, ε, ενός γενικότερου ε, προβληματισμού για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Να υπενθυμίσω λοιπόν καταρχήν ότι η Κομισιόν και το Συμβούλιο και το Συμβούλιο πέρυσι δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν για την παράταση για την οποία συζητάμε σήμερα. Λόγω του ότι αυτή η πρόταση συζητήθηκε στα πλαίσια των παλιών διαδικασιών πριν από την ε, εφαρμογή της συνθήκης της ε, Λισαβόνας. Σήμερα τώρα οι διαδικασίες της συνθήκης Λισαβόνας ισχύουν και μια νέα παράταση του κανονισμού περνάει μέσω ενός διαλόγου και μάλιστα τριμερούς διαλόγου αρκετά ενδελεχούς. Το πλαίσιο της παράτασης βασίζεται στην ανάγκη να κάνουμε μια αξιολόγηση επιπτώσεων των μέτρων αυτών στον τομέα της αλίας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2013. Ακριβώς την ημερομηνία για την οποία προβλέπουμε την παράταση του μηχανισμού αυτού. Τώρα ο μηχανισμός αυτός καθεαυτός που έχετε μπροστά σας αντιγράφει αυτά που υπήρχαν μέχρι πέρυσι και απλώς παρατείνονται. Θέλουμε δηλαδή να ισχύσουν τα ίδια μέτρα που υπήρχαν στον μηχανισμό των ΤΑΚ και ποσοστώσεων και με βάση και επίσης ποια μέτρα δεν μπορούσαν να παραταθούν ε, με βάση το άρθρο 43.3 της συνθήκης. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν εξετάζουμε αυτή την παράταση. Η συγκήτρια μας ρώτησε ποιες είναι οι προθέσεις μας στα πλαίσια της μεταρρύθμισης. Καταλαβαίνετε ότι επειδή η ημερομηνία της παράτασης και η ημερομηνία εφαρμογή τη μεταρρύθμιση κοινή αλληλευτική πολιτική συμπίπτων, μπορεί να έχουμε ένα κεφάλαιο για τα τεχνικά μέτρα στον βασικό κανονισμό τη μεταρρύθμιση που θα, έχει τα ουσιαστικά, θα περιλαμβάνει τα ουσιαστικά μέτρα για την εφαρμογή τη ε, συνθήκη σε τεχνικό επίπεδο και εν συνεχεία η Κομισιόν σύμφωνα με την προηγούμενη πρότασή της θα θελήσει να, να τα εφαρμόσει περιφερειακά μέσω ε, πράξεων κατεξουσιοδότηση ή μέτρων κατεξουσιοδότηση. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Όλα αυτά θα τα δούμε στα πλαίσια του πακέτου της μεταρρύθμισης. Προς το παρόν ζητάμε να μας εγκρίνεται απλώς την παράταση του σημερινού καθεστώτος. Τίποτα περισσότερο. Πολύ ωραία. Ο κύριος Γκάλαχερ. Μπορεί να φαίνεται πολύ απλό αυτό το αίτημα να το επεκτείνουμε, αλλά μήπως πρέπει να δούμε λίγο και το κατά πόσο είναι πρακτικό αυτό, γιατί το Συμβούλιο και η Κομισιόν δεν συμφώνησαν επ' αυτό. Αυτό που περιλαμβάνεται εδώ είναι αυτό που λέμε εδώ και καιρό και συνεχώς ότι έχουμε έναν ε, κανόνα και, το ένα, και μια πανάκια ένα μέτρο για όλους. Ελπίζω το 2013 να έχουμε κάποια μέτρα που θα περιλαμβάνουν μέτρα και για την κοινή ε, πολιτική αλίας. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πουλήσουμε καλά αυτά. Ας πούμε, πάρτε ένα 15 μέτρο σκάφος κάποια κουτιά είπαμε ότι δεν, κάποια σκάφη μάλλον σε, κάποια, ε, σε κάποιες περιφέρειες είπαμε ότι δεν θα αλλιεύουν. Και κάποια ε, σκάφη θα πρέπει υποχρεωτικά να ταξιδεύουν ε, πέρα από αυτές τις ζώνες για 4, 5, 6 ώρες για να αλλιεύσουν. Οπότε οι επιπτώσεις για αυτούς που θα μπορούσαν να έχουν εισόδημα πιο κοντά στο δικό τους λιμάνι από το να ταξιδεύουν 5-6 ε, ώρες θα ήταν μεγαλύτερο. Και νομίζω ότι γι' αυτό θα φταίμε εμείς αν τελικά γίνει. Θα φταίμε εμείς για τους κινδύνους που θα, που θα έχουν να αντιμετωπίσουν αυτοί οι άνθρωποι για να ταξιδέψουν 5 ώρες για να έχουν εισόδημα και να μπορέσουν να ξεπληρώσουν τις τράπεζες. Το έχουμε πει πολλές φορές εδώ. Οι επιπτώσεις ε, που, ε, που έχουν οι κανόνες αυτοί σε μικρά σκάφη και στα συνολικά αλλιεύματα είναι πραγματικά ε, πολύ μικρές. Γι' αυτό ο κανόνας αυτός θα πρέπει να ισχύει για όλους. Είτε είναι το σκάφος 15 μέτρα είτε είναι 115 μέτρα. Το είχαμε πει ήδη και στο Λουξεμβούργο από το 2009, έτσι ώστε να καταλέξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Ότι δηλαδή είπαμε ότι θα υπάρχουν κάποιε συγκεκριμένε προτάσει. Και τώρα τι λέμε, λέμε ότι θα παραμείνει η κατάσταση έτσι για άλλο ένα μισή χρόνο. Ε, ναι, αλλά εντάξει, εκ πρώτη όψεω φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο λογικό επιχείρημα για να υπάρξει αυτό το αίτημα, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει τελικά αυτό. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω, θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη επαφή με την Κομισιόν και όντω με τα γνωμοδοτικά συμβούλια, τα περιφερειακά, για να δούμε ποιε είναι οι επιπτώσει. Δεν ξέρω βέβαια πώ έχει η ατζέντα τη Επιτροπή μα, αλλά νομίζω ότι ένα από τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια θα πρέπει να ζητηθεί να στείλει έναν ε, εκπρόσωπό του και να μα πει ποιε είναι οι επιπτώσει αυτών των κανόνων ε, ε, βραχυπρόθεσμα. Πρόεδρε, δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα να συμφωνήσω με την επέκταση των μέτρων αυτών μέχρι τον επόμενο Ιούνιο, εάν αυτό είναι απαραίτητο, γιατί αλλιώς θα εκπνεύσουν. Το θέμα είναι μετά τον Ιούνιο τι γίνεται. Γιατί ήδη αυτό το έχουμε συζητήσει και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Αν δηλαδή η πρόθεση της Κομισιόν να, να παράγει αυτό το πλαίσιο και να έχει αυτό το τεχνικό λεπτομερές ντοσιέ με όλα τα μέτρα είναι ε, σωστό. Ε, αυτό το πλαίσιο αυτό που θα, για την περιφερειοποίηση που θα υποβάλλεται σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθούν, θα μεταφερθούν δηλαδή αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες στις περιφέρειες κατευθείαν ή θα υπάρξει επιτροπολογία. Γιατί εκεί είναι πάντα ο διάβολος, τη λεπτομέρεια. Αν υπάρξει επιτροπολογία θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Αν δηλαδή πάμε στις περιφέρειες και τους ε, ε δώσουμε εμείς ε, λεπτομέρειες ε, ε, για τις δικές τους δραστηριότητες, εντάξει, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια της γενικότερης κοινής ελευτικής πολιτικής. Λοιπόν, ελπίζω να μην μπούμε στην επιτροπολογία, γιατί έτσι έγινε εφικτό να μπλοκάρει το θέμα το Συμβούλιο. Φαντάζομαι λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα επιλέξει την επιτροπολογία στο μέλλον. Έχετε το λόγο, εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να απαντήσω στον κύριο Γκάλαγκερ, για τις ανησυχίες που έχει σε ό,τι αφορά τη σημερινή κατάσταση. Για τα σκάφη και ιδίως τα μικρά σκάφη με βάση τα σημερινά, τα όσα ισχύουν σήμερα. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε να εκπνεύσει το σημερινό σύστημα για να γίνει μια αξιολόγηση επιπτώσεων για να καταλάβουμε πού αποτύχαμε τον περασμένο Νοέμβριο ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι για να αναπτύξουμε καλύτερα μέτρα που ευθυγραμμίζονται περισσότερο και λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες του κλάδου. Δηλαδή, επειδή παρατείνουμε κάποια μέτρα, δεν σημαίνει ότι σταυρώνουμε και τα χέρια στο μεταξύ. Μπορείτε να μου πείτε, ας αναπτύξουμε αυτά τα μέτρα πάρα αυτά. Αλλά αυτό δεν είναι ευκταίο γιατί θα είμαστε εκτός πλαισίου της μεταρρύθμισης. Αντίθετα, θα πρέπει και εσείς να ανησυχείτε, όπως και εμείς ανησυχούμε, για το θέμα της αξιολόγησης ε, των επιπτώσεων. Για τα μέτρα που ήδη συζητώνται. Αυτή η πρόταση παράτασης συζητείται στο Συμβούλιο και εμείς έχουμε κάποια αιτήματα ε, από κράτη-μέλη που θέλουν βελτιώσεις στο σημερινό σύστημα. Ε, βελτιώσεις που τις γνωρίζουμε και που ε, αξιολογούνται από τους αρμόδιους επιστημονικούς οργανισμούς. Είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε παράλληλα σε αυτήν την περίοδο παράτασης ένα νέο καθεστώς τεχνικών μέτρων που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στη σημερινή πραγματικότητα της, ε, των αλληλευτικών δραστηριοτήτων. Τώρα, ποιες είναι οι διαδικασίες μέσω των οποίων ε, υιοθετούμε αυτό το νέο καθεστώς δεν μπορώ να πω εδώ για το ποιο. Γιατί εδώ έχει να κάνει με το, περι... περιεχόμενο της ε, μεταρρύθμιση για την περιφερειοποίηση. Αυτό ακόμα συζητείτε. Σε ποιο βαθμό η εφαρμογή εφαρμοστικών μέτρων της μεταρρύθμισης θα γίνει μέσω της επιτροπολογίας, μέσω της περιφερειοποίησης που θα είναι εκτεταμένη λιγότερο ή περισσότερο μέσω μηχανισμών που εφαρμόζουν απευθείας τα κράτη-μέλη, τι να σας πω, δεν μπορώ να σας απαντήσω σήμερα όπως και εσείς ε, δεν ξέρετε, παρότι έχω καθένα στις ιδέες του δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η Κομισιόν θέλει μια περιφερειοποίηση. Δηλαδή, μια εφαρμογή περιφερειακή των τεχνικών μέτρων. Με βάση το βαθμό εκμετάλλευσης, με βάση τη φύση των αποθεμάτων και με βάση το, την κατάσταση του αλευτικού στόλου, που είναι μεικτός και που δημιουργεί προβλήματα σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση. Non, je marqué, euh, Monsieur le Président la Commission, qu'il vient répondre à la question que j'avais tenté de lui poser. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ε, κρατήστε μας ενήμερους για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ε, στο μεταξύ μας είπατε ότι θα σκεφτείτε ε, για τη δυνατότητα ενός νέου καθεστώτος. Ενημερώστε μας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αποτυχίες. Ε, το θέμα αυτό πάντως είναι επιτάπητος επί 2008. Φαντάζομαι ότι έχετε διάφορες προθέσεις. οι προθέσεις αυτές βέβαια εντάσσονται ε, στα πλαίσια της ε, μελλοντικής μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Καλώς. Λοιπόν, στη συνεδρίαση της 30 Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί η έκθεση αυτή. Περνάμε στο σημείο 12. Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή μετά τη λήξη των εξαιρέσεων από την εφαρμογή ορισμένων τεχνικών μέτρων στην Μεσόγειο. Η αρμόδια εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει έρθει ακόμα. Να περιμένουμε 5 λεπτά. Διακόπτουμε τη συνεδρίαση για 5 λεπτά να επιστρέψετε όμως, κυρίως όσοι έχετε ζητήσει να λάβει χώρα τέτοιου είδους συζήτηση. Σε πέντε λεπτά να επιστρέψετε όλοι παρακαλώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αλίας. Είμαστε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τη λήξη των εξαιρέσεων από την εφαρμογή ορισμένων τεχνικών μέτρων στην Μεσόγειο. Το συζητήσαμε το θέμα αυτό μία φορά πριν από κάποιους μήνες και μετά από αίτημα της ομάδας των Πρασίνων το ξανασυζητούμε και σήμερα διότι αν δεν απατώμε στην τελευταία συνοδρίαση ε, υπόθηκε ότι ορισμένα κράτη δεν έχουν ακόμα υποβάλει σχέδια διαχείρισης, άρα καλό θα ήταν να μας ενημερώσει η Επιτροπή για το πώς έχει η κατάσταση, αν έχουν υποβληθεί όλα τα σχέδια διαχείρισης και βεβαίως θα πρέπει αυτά να συμμορφώνονται με τον κανονισμό για τα τεχνικά μέτρα. Είναι νωρίς βέβαια ακόμα, αλλά αν έχετε άποψη και γνώση για τον βαθμό στον οποίο έχουν εκπληρώσει τα κράτη τις ε, υποχρεώσεις τους, καλό θα είναι να το μοιραστείτε μαζί μας. Καλωσορίζω την κυρία Τάρια, αν προφέρω σωστά το όνομά της, πρώην ε, υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Αλίας, η οποία πλέον έχει επιστρέψει στην καινούργια Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων. Μάρε, καλωσορίζουμε λοιπόν την εκπρόσωπο στη δική μας Επιτροπή Αλληλείας. Το γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα αυτό, είναι πολύ σημαντικό, ενδιαφέρει πολλά μέλη του Κοινοβουλίου, είμαστε λίγοι εδώ παρόντες, ωστόσο θα διαβιβάσουμε τις πληροφορίες και στους υπόλοιπους και μας ενδιαφέρει ε, το πώς εξελίσσεται ο κανονισμός αυτός για τα τεχνικά μέτρα. Σας δίνω ευθύς αμέσως το λόγο για να μας ενημερώσετε. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τα καλά σας λόγια επίσης. Να σας εξηγήσω ποια είναι η κατάσταση για τον κανονισμό για τη Μεσόγειο. Χαίρομαι που ζητήσατε αυτή τη συνάντηση, γιατί μας δίνετε την ευκαιρία να σε για την ε, εφαρμογή του κανονισμού για τη Μεσόγειο μετά από τη συνάντηση που είχαμε τον Ιούλιο, στην οποία αναφερθήκατε. Ο κανονισμό αυτός, όπως γνωρίζετε, είναι περίπλοκος και πολύ ευρύς και καλύπτει όλα τα είδη αλίας και έχει και περιβαλλοντικά μέτρα που περιλαμβάνονται στις τομεακές πολιτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Μεσογειακής Λεκάνης είναι καρπός μιας μεγάλης ε, διαδικασίας ε, διαπραγμάτευσης. Δεν, ήταν, δεν θα είναι εύκολος ο ε, κανονισμός για να εφαρμοστεί και τα κράτη-μέλη έχουν δείξει ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους κατά την εφαρμογή του κανονισμού. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να κατανοήσουν καλύτερα τον κανονισμό και να υλοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους με τη δημιουργία του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού, Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Μεσόγειο που έγινε λειτουργικό το 2010. Η Κομισιόν ε, συμμετείχε σε διάφορες ε, συναντήσεις στη Μαρμπέγια και στη Θεσσαλονίκη για να δώσει κάποιες εξηγήσεις για διάφορα θέματα. Επίσης ε, έγιναν και άλλες ε, Επαφέ της Κομισιόν με διάφορους ενδιαφερόμενους για τη Μεσόγειο σε διάφορες συναντήσεις για να δώσουμε πληροφορίε και να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Η κυρία Δαμανάκη, Επίτροπο, πήγε στην Ελλάδα για να συναντήσει διάφορες οργανώσει αλλιέων και μη κυβερνητικές οργανώσει. για να βοηθήσει τον τομέα της αλίας. και, τα, και τους διαχειριστικούς φορείς. Τα κράτη-μέλη προέβησαν σε αναθεώρηση των εθνικών διαχειριστικών προγραμμάτων, τα οποία γνωρίζετε ότι στηρίζουν ε, τα αιτήματά τους για παρεκκλήσεις. Θα γνωρίζετε ίσως ότι υπάρχει υποχρέωση να συντάξουν τα κράτη-μέλη εθνικά διαχειριστικά προγράμματα για όλα τα αλλιεύματα και αν ζητάνε παρέκκληση, ο κανονισμός προβλέπει ότι θα πρέπει να γίνει με βάση ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης. Θα πρέπει δηλαδή αυτή η παρέκκληση να δοθεί μόνο υπό αυτού του όρου. Υπάρχουν διάφορε διαδικασίε, δεν θα αναφερθώ, δεν θα αναφερθώ σε αυτέ, αλλά μπορώ να επανέλθω αν θέλετε. Οι διαδικασίε λένε ότι μόνο σε περίπτωση που ζητούνται παρεκκλήσεις χρειάζονται εθνικά διαχειριστικά μέτρα. Παραδείγματο χάρη παρεκκλήσεις από την απόσταση από την ακτογραμμή. Υπάρχουν διαδικασίες, ζητείται η γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής και τότε θα πρέπει να πάμε στη διαδικασία της επιτροπολογίας. Εντό αν άμα επιτρέπετε τον όρο, επιτροπολογία. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι ο κανονισμός για τη Μεσόγειο υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2006 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2007. Τα κράτη-μέλη είχαν μέχρι το Δεκέμβριο του 2007 για να υποβάλουν και να υιοθετήσουν τα εθνικά προγράμματα ή σχέδια διαχείρισης. Ξέρω ότι τα περισσότερα δεν το έκαναν. Και τελικά Λάβαμε κάποια από αυτά τα σχέδια μεταξύ του 2007 και της σημερινής ημέρας, αλλά υπήρχαν ελλείψεις στις πληροφορίες ή υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις που δεν είχαν γίνει σεβαστές, γι' αυτό ζητούσαμε περαιτέρω πληροφορίες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι στο τέλος του Μαΐου του 2010, όπου η προθεσμία για τις παρεκκλήσεις κανονικά εξέπνε, δεν υπήρχε κανένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης για παρεκκλήσεις ή που θα επέτρεπε τις παρεκκλήσεις. Επομένως, το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι δεν έχει δοθεί καμία παρέκκληση. Γιατί δεν είχαμε κανένα ισχύον σχέδιο διαχείρισης. Δηλαδή κανένα σχέδιο που να έχει όλες τι απαραίτητες πληροφορίες που θα έπρεπε να διαβιβαστούν στην Επιστημονική Επιτροπή και συνεχεία να πάνε στη διαδικασία της επιτροπολογίας όπως προβλέπετε. Ή κανένα τέτοιο σχέδιο, προς εθνικό σχέδιο διαχείρισης, επί του οποίου θα μπορούσαμε κατευθείαν να πούμε εντάξει, να συμφωνήσουμε αμέσως. Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Ιουνίου του 2010 δεν έχει χορηγηθεί καμία παρέκκληση. Καμία παρέκκληση δεν μπορεί να χορηγηθεί, καμία παρέκκληση δεν γίνεται δεκτή για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού για τη Μεσόγειο. Επίσης, λάβαμε κάποια διαχειριστικά σχέδια λίγο πριν την εκπνοή τη προθεσμία, 27 Μαΐου, 28 Μαΐου, τότε λάβαμε τα περισσότερα. Καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε χρόνο για να τα εξετάσουμε. Χρειαζόμαστε χρόνο για να αναλύσουμε το κατά πόσον ισχύουν με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στα παραρτήματα του κανονισμού. Εν συνεχεία έπρεπε να περάσουμε από την Επιστημονική Επιτροπή και μέχρι στιγμής έχουμε μόνο δύο σχέδια που θα περάσουν από την Επιστημονική Επιτροπή τον Νοέμβριο, ένα της Ισπανίας και ένα της Ιταλίας. Και αναλόγως με το τι θα αποφανθεί η Επιστημονική Επιτροπή και ανάλογα με το τι θα προκύψει από τη δική μας ανάλυση, εν συνεχεία θα περάσουμε από τη Διαχειριστική Επιτροπή με την ελπίδα ότι θα τα υιοθετήσουμε στις αρχές του 2011. Η κατάσταση δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Αλλά έχουμε σχέδια διαχείρισης αυτή τη στιγμή τώρα για εννέα Είναι υπό εξέταση, όπως σας είπα. Αποφασίσαμε επίσης να έχουμε τακτικές επαφές με τα κράτη-μέλη για να επιταχύνουμε όσο μπορούμε τις διαδικασίες και να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με τα κράτη-μέλη και τη διοίκησή τους για να διευκρινίσουμε τα σκοτεινά σημεία αυτών των σχεδίων διαχείρισης με σκοπό να τα υιοθετήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Αυτά έτσι σε αδρέ γραμμές μπορώ να επανέλθω σε πιο τεχνικά σημεία, να μπω σε λεπτομέρειε, να σχολιάσω τα σχέδια αυτά των εθνικών, τα επιμέρους σχέδια των κρατών μελών, αλλά σε αδρές γραμμές αυτή είναι η κατάσταση. Ευχαριστώ, κυρία Λαβίν. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για αυτές τις πολύ ξεκάθαρες εξηγήσεις. Βεβαίω, τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να υποβάλουν ε, σχέδια διαχείρισης ακόμα, ενώ η απόφαση έχει ληφθεί για αυτά από το Δεκέμβριο του 2006 και βεβαίως αυτό μας βρίσκει αντίθετους και το επικρίνουμε ιδιαιτέρως ως ε, στάση. Πόσες παρεκκλήσεις ζητήθηκαν, είπατε ότι καμία δεν δόθηκε. Πόσες όμως ζητήθηκαν, αυτό είναι το ερώτημά μας. Και άλλο ερώτημα είναι το εξής. Έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια από τα σχέδια διαχείρισης που έχει υποβάλει κάποιο κράτος μέλος ή συνεχίζει να τα εξετάζει όλα χωρίς να έχει εγκρίνει κάποιο οριστικά. Αυτά είναι τα ερωτήματά μου. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, η κυρία Αντρές Παρέα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω ένα διευκρινιστικό ερώτημα. Η Ιταλία και η Ισπανία έχουν υποβάλει σχέδια διαχείρισης, τα οποία θα εξετάσει τώρα η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα εκδώσει μια γνωμοδότηση και θα κάνει την αξιολόγηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιο είναι το επόμενο βήμα θα πρέπει το κράτος μέλος να προσαρμόσει τα πεπραγμένα εάν δεν πληρεί βάση της Επιστημονικής Επιτροπής κάποιο από κάποια από τις προϋποθέσεις για να πάει μετά το θέμα στην Επιτροπολογία. Ποιο είναι το επόμενο στάδιο δηλαδή είναι το ερώτημα. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Για το πρώτο ερώτημα που μου θέσατε. Όπως είπα και προηγουμένως, νέα κράτη-μέλη ζήτησαν παρεκκλήσεις ως προς την απόσταση από τα παράλια. Ε, και αυτή είναι και η πιο σημαντική παρέκκληση βεβαίως βάσει του κανονισμού. Μιλούμε για το άρθρο 13.5.9. 9 κράτη-μέλη λοιπόν. Όχι, διορθώνω λέει η ομιλήτρια. 7 ε, κράτη-μέλη. Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα και Σλοβανία πέντε, μας ανέφερε η ομιλήτρια. Αυτά τα κράτη-μέλη ζήτησαν παρέκκληση. Η Ιταλία έχει εγκρίνει οκτώ σχέδια διαχείρισης ήδη, χωρίς όμως παρεκκλήσεις. Είναι σχέδια χωρίς καμία παρέκκληση. Όπως σας εξήγησα και προηγουμένως, επαναλαμβάνω τη διαδικασία. Ένα κράτος μέλος καταρτίζει ένα σχέδιο διαχείρισης, στη συνέχεια το υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον έξι μήνες πριν προχωρήσει στην έγκρισή του, ώστε να έχει χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφανθεί επ' αυτού του σχεδίου διαχείρισης. Αυτό έγινε και με την Ιταλία. Τα σχέδια λοιπόν που δεν προέβλεπαν παρεκκλήσεις τα Ιταλικά εγκρίθηκαν και έγιναν μέρος της Ιταλικής νομοθεσίας. Βεβαίως εξετάζουμε ε, το κατά πόσο οι τροποποιήσεις που ζήτησαμε από την Ιταλία ε, να κάνει, εάν τις έχει κάνει και αν έχει προβεί σε αυτές. Εν πάση περιπτώσει, τα σχέδια αυτά έχουν εγκριθεί έχουν ενσωματωθεί στην Ιταλική ένομη τάξη. Τώρα, ως προς το δεύτερο ερώτημα, όταν λαμβάνουμε ένα σχέδιο διαχείρισης, τι κάνουμε πρώτα απ' όλα. Επιβεβαιώνουμε ότι έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία που ζητούμε. Ε, χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα κριτήρια. Ιδαλλιώς δεν το στέλνουμε το σχέδιο αυτό στην Επιστημονική Επιτροπή, το επιστρέφουμε στο κράτος μέλος. Εάν λοιπόν εξετάσουμε το σχέδιο διαχείρισης και δούμε ότι όντως περιλαμβάνει τα στοιχεία που ζητήσαμε, τότε το στέλνουμε στην Επιστημονική Επιτροπή. Δύο είναι τώρα οι εναλλακτικέ. Η Επιστημονική Επιτροπή μπορεί να πει καλώς δεν υπάρχει τίποτα εδώ το περίεργο, άρα ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρούμε στην ανάλυση μας και το καθεξής και στη συνέχεια πάει το θέμα στη διαχειριστική επιτροπή. Εάν η επιστημονική επιτροπή δεν καλυφθεί και ζητήσει περισσότερα στοιχεία, τα ζητάει από εμά, τα διαβιβάζουμε εμεί στο κράτο μέλο, διαβιβάζουμε το ερώτημα, δηλαδή το έτοιμο τη επιστημονική επιτροπή και κάνουμε αυτή τη δουλειά τη παρακολούθηση ώστε να μα επιστρέψει το κράτο μέλο τα στοιχεία που δεν είχε υποβάλει αρχικά για να τα υποβάλουμε στην επιστημονική επιτροπή και να ε, καλυφθεί. Άρα εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διασφαλίζουμε ότι έχει ολοκληρωθεί κάθε στάδιο σωστά. Πρώτον, ότι είναι ευανάγνωστο το σχέδιο, δηλαδή περιλαμβάνει τα στοιχεία που χρειάζεται. Εάν ναι, το στέλνουμε στην Επιστημονική Επιτροπή, καλύπτεται αυτή. Αν δεν καλύπτεται, ξαναζητούμε ε, αυτά που λείπουν από το κράτος μέλος. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το εξής σε περίπτωση κατά την οποία δεν μας ικανοποιεί καθόλου το σχέδιο διαχείρισης που προτείνει το κράτος μέλος, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμείς έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε σε επίπεδο Επιτροπής ένα διαχειριστικό σχέδιο λευκό, όπως λέει η ομιλήτρια δεν είναι μια άγουσα την οποία έχουμε ακολουθήσει. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι τέτοιο για να αποφύγουμε την κακή διαχείριση της αλληλείας από το λόγο κράτος μέλος. Δεν έχει συμβεί ακόμα, δεν το έχουμε κάνει. Μέχρι στιγμής συνεργαζόμαστε εκ του σύνοικης με τα κράτη-μέλη για να έχουμε εθνικά διαχειριστικά σχέδια για τη σωστή διαχείριση των αλληλευτικών πόρων. Η κυρία Μπάρια. Βαρέα. Ναι, ένα διευκρινιστικό ερώτημα. Εννέα κράτη-μέλη είπατε ότι έχουν υποβάλει σχέδια διαχείρισης. Δύο έχουν περάσει και από την Επιστημονική Επιτροπή, το Ιταλικό και το Ισπανικό, και επτά ε, ακόμα δεν έχουν περάσει από την Επιστημονική Επιτροπή και τίθεται το θέμα της παρέκκλησης από την, ως προς την απόσταση από τα παράκτια. Ε, με ποια βάση ε, κάνουν αυτό το αίτημα, μπορείτε να μου το διευκρινίσετε, πού ε, ακριβώς το στηρίζουν η Πρόεδρο. Σας υπενθυμίζω ότι το άρθρο 13 δίνει δυνατότητε παρέκκληση από τα παράκτια βάσει τη γεωμορφολογία του εδάφου και ούτω υπό τον όρο ότι θα τεκμηριωθούν επιστημονικώ και Να δώσουμε το ίδιο μέτρο σε όλε τι ζώνε, σε όλε τι περιοχέ ανεξαρτήτως γεωμορφολογίας είναι κάτι το πολύ δύσκολο και πολύ περίπλοκο. Επομένω, αναλόγω με ορισμένε παραμέτρου, και αν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση από αυτού και κάθε φορά που υποβάλλεται ένα σχέδιο διαχείριση, τότε μπορεί να ε, δοθεί λαβή, να υπάρχει δηλαδή νομική βάση για παρέκκληση και ούτω καθεξής. Αυτά λέει εν συντομία το άρθρο 13 και είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί επανειλημμένως. Εγώ είχα διαπραγματευτεί για το θέμα αυτό και γι' αυτό τα θυμάμαι τόσο καλά. Να κάνω κάποια σχόλια όμω και δεν θέλω να επικρίνω καθόλου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτού, ωστόσο να επικρίνω την κατάσταση που επικρατεί στη Μεσόγειο αυτή τη στιγμή. Και το μόνο που λέω είναι ότι εάν τα διαχειριστικά σχέδια πρέπει να υποβάλλονται σε συγκεκριμένη προθεσμία και δεν γίνεται, δεν γίνεται κάτι τέτοιο, ε, δεν θα πρέπει να υπάρξει κάποια κύρωση για το λόγο Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει για να μην ε, γίνει ε, ανεκδοτική κατάσταση στη Μεσόγειο. Ε, ο κλάδος δεν θέλει να υποβάλει τέτοια πράγματα και δεν θέλει να συμμορφούνται με τον κανονισμό με τα τεχνικά μέτρα. Δεν ξέρω όμως τι συμβαίνει με το κάθε κράτος μέλος. Το κράτος μέλος όμως δεν συνεργάζεται. Όταν ο κράτος δεν το επιθυμεί, το, κλάδο, το κράτος δεν συνεργάζεται, δεν υποβάλλει σχέδια διαχείρισης. Έχουμε δυνατότητες παρεκκλήσεων. Τεκμηριωμένες. Επομένως θα πρέπει να υποβάλλονται σχέδια διαχείρισης. Όταν δεν υποβάλλονται θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες κυρώσεις. Ο κλάδος έρχεται και διαμαρτύρεται και, το... και δικαίως αν θέλετε γιατί ούτε το κράτος μέλος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις τους. Εδώ δεν έχουμε βουλευτές από την Ιταλία, όμως η... Α, έχουμε, συγγνώμη, δεν σας είχα δει. Αλλά ε, είναι αλήθεια αυτό που λέω. Έρχονται οι Ιταλοί αλληλεί και παραπονιούνται συνεχώ, παραπονιούνται συνεχώς και ε, η Ιταλική κυβέρνηση δεν έχει υποβάλει ακόμα σχέδιο διαχείριση. Δεν είστε μέλος της ε, υφιστάμενης κυβέρνηση στην Ιταλία. Επομένω, δεν σα αφορά και δεν σα νοιάζει που επικρίνω τόσο πολύ την Ιταλική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν έχουν υποβάλει σχέδια διαχείρισης και αν υποβάλουν σχέδια διαχείρισης οι Ιταλοί δεν ζητούν παρεκκλήσεις ενώ τις θέλει ο Ιταλικός κλάδος και τις ζητούν οι Ιταλοί αλληλείς. Δηλαδή είναι λίγο κοροϊδία. Κανείς δεν θέλει να κάνει τίποτα για τη Μεσόγειο. Θα μου άρεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το θέσει το θέμα με σοβαρότητα στα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη. Από το 2006 μέχρι σήμερα δεν έχουμε σημειώσει καμία πρόοδο και δεν ξέρω γιατί έχουμε κανονισμό εάν δεν τον εφαρμόζει κανείς. Έχω πάω, εγώ έχω πάει πολλές φορές και στην Ισπανία και στην Ιταλία και όλοι μου λένε «Μα δεν θα τον τηρήσουμε τον κανονισμό, δεν θα τον εφαρμόσουμε, είναι καταστροφική η κατάσταση». Τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια το ίδιο. Το μοναδικό περιφερειακό γνωμοδοτικό συμβούλιο στο οποίο δεν πιστεύουν τα μέλη του είναι αυτό της Μεσογείου, σε όλο τον κόσμο. Ίσως θα έπρεπε κάτι να κάνουμε πραγματικά. Αλλιώς ε, να πετάξουμε λευκή πετσέτα και να παρετηθούμε. Ο παλιότερος κανονισμός δεν το και δεν εφαρμοζόταν διότι ήταν τελείως παράλογος και αντιφατικός δεν ε, είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο τωρινός κανονισμός είναι αρκετά λογικός, δηλαδή έγινε προσπάθεια να ε, εκλογικευτεί η κατάσταση, αλλά ούτε αυτός εφαρμόζεται, ούτε αυτό στηρείται, κανένα από τα μέλη δεν θέλει να τον τηρήσει και να τον εφαρμόσει. Έχετε κάποια ιδέα, εσείς Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποιο μέλος του Κοινοβουλίου, έχει κάποια ιδέα για το πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλιώς συζητούμε επί μακρόν, ε, το έχουμε κουράσει το θέμα χωρίς να έχουμε προχωρήσει. Τι θα γίνει στη Μεσόγειο, δηλαδή να τα αφήσουμε όλα στο έλεος του Θεού, μήπως γίνει κάτι ή μπορούμε κάπου να δράσουμε, μπορούμε κάτι να κάνουμε και είναι κάτι που πραγματικά με πονάει γιατί εγώ μαζί με άλλους ανθρώπους έχουμε δουλέψει πραγματικά ε, για να βελτιωθεί η κατάσταση και δεν γίνεται τίποτα. Καταλαβαίνω την απόγνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάνω αυτές τις γενικές παρατηρήσεις και τα γενικά σχόλια και αν έχει κάποιος κάποια ιδέα για να μας διαφωτίσει είναι ευπρόσδεκτη η ιδέα αυτή. Μήπως μπορούμε να ε, αλλάξουμε το ρου ε, των πραγμάτων, αλλιώς να το ξεχάσουμε. Κυρία Λέβιν, παρακαλώ. Well, yes, actually we have an idea. If we all... Ναι, αλλά Πρόεδρε, εφόσον όλοι ε, ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε μια κοινή ελληνική πολιτική και ένα κομμάτι αυτής της πολιτικής είναι να υπάρχει ένα ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αλληλεία, θεωρώ ότι τα κρατη που δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προφανή τρόπο δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ίσως θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη τα οποία δεν συμμορφώνονται δεν λαμβάνουν βοήθεια. Αυτό προβλέπεται και στο βασικό κανονισμό. Ε, ίδιες αρχές που ισχύουν σε όλες τις συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, για όλα τα θέματα. Όποιος δεν συμμορφώνεται πληρώνει. Κομισιόν, εσείς μπορείτε να μας διαφωτίσετε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτήν την κατάσταση, ε, έστω λίγο. Εσείς αντιμετωπίζετε τώρα και τον κλάδο. Απ' τη μία έχετε τον κλάδο, από την άλλη έχετε τα κράτη-μέλη. Έχετε αυτά τα σχέδια διαχείρισης μπροστά σας, τα οποία θα πρέπει να επικυρωθούν τελικά από την ε, Επιστημονική Επιτροπή. Ε, μπορείτε να μας βοηθήσετε εμείς που πλέουμε μέσα σε πελάγια απογοήτευσης. Ευχαριστώ κυρία Φράγκα. Ξεκίνησα με τα θετικά των δράσεών μας. Υπάρχουν και τα αρνητικά. Ας πούμε ο έλεγχος και η συμμόρφωση και η εποπτεία η συμμόρφωση με τους κανονισμούς, οι διαδικασίες επί παραβάση που μπορούμε να ξεκινήσουμε. Οπότε, από τη μια δείχνουμε μεγάλη υπομονή με τα κράτη-μέλη και κατανοήσαμε ότι αυτός ο κανονισμός δεν είναι εύκολος για να εφαρμοστεί, αλλά ε, όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο. Οπότε εμεί προσπαθούμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας έτσι ώστε τα διαχειριστικά σχέδια που έχουμε τώρα θα περάσουν το δυνατόν συντομότερο και ταυτόχρονα Θέλουμε να έχουμε ένα αυστηρό πρόγραμμα ελέγχου για τη Μεσόγειο όπως και για άλλες, άλλα σημεία του πλανήτη όπου θέλουμε ε, όπου παρατηρούμε ποια είναι η ε, διαδικασία που παραβιάζεται και πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε την σχετική ε, διαδικασία. Με βάση όμως αυτόν τον κανονισμό θα μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες επί παραβάση. Η Κομισιόν είναι σαφέστατη ως προς αυτό και θέλει να εφαρμοστεί ο κανονισμός. Οπότε στην φαρέτρα των όπλων μας θα έχουμε άλλο ένα, αυτό το κανονισμό. Και θα ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τα διαχειριστικά προγράμματα. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αποφασίσουμε ότι θα υπάρχει διαχειριστικό σχέδιο ευρωπαϊκό. Παράλληλα, θα φροντίσουμε όσο μας επιτρέπουν τα μέσα που έχουμε να έχουμε και έναν ε, ενδελεχή έλεγχο της κατάστασης. Ήδη έχουμε κάνει κάποιους, κάποιους ελέγχους σε κάποια κρατημέλη όπου η κατάσταση δεν είναι απολύτως ικανοποιητική και εξακολουθούμε να έχουμε την, το δικαίωμα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία επί παραβάση. Ο κανονισμός ελέγχου μας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε και μια ε, διοικητική έρευνα για το πώς διαχειρίζεται κανείς την αλληλεία. Αυτή είναι άλλη μια δυνατότητα που έχουμε και επίσης ε, μελετούμε προγράμματα εποπτείας από κοινού με την ε, υπηρεσία ελέγχου, την κοινωτική υπηρεσία ελέγχου αλίας, Οπότε δουλεύουμε και στα δύο μέτωπα. Συνεργασία μεν με τα κράτη-μέλη, αλλά και εφαρμογή αυστηρού, αυστηρής πολιτικής ελέγχου και συμμόρφωσης. Και ως προς αυτό θα χρησιμοποιήσουμε όλα μας τα μέσα, ώστε να εφαρμοστεί στο ακέραιο αυτός ο κανονισμός. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι και καινή ώρα να ξεκινήσει κάποια πειθαρχική διαδικασία, κάποια διαδικασία επί παραβάση. Τουλάχιστον για ένα κράτος μέλος. Νομίζω ότι η έλλειψη της συμμόρφωσης είναι γενικευμένη. Εγώ μίλησα απλώς με τους εκπροσώπους του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Αυτοί μου λένε ότι με αυτόν τον κανονισμό. Κανένας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλοι το ξέρουμε. Ο καθένας έχει τις ευθύνες του αφού το ξέρουμε. Και τα κράτη-μέλη βεβαίως έχουν τις περισσότερες ευθύνες. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν σέβεται κανένας τον κανονισμό. Ε, ίσως κάποιοι συμμορφώνονται μερικώς, αλλά κανένας δεν συμμορφώνεται πλήρως με αυτόν τον κανονισμό. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Ε, δεν άλλαξε τίποτα από την τελευταία φορά που τα είπαμε για το θέμα αυτό. Χαίρομαι όμως που ήρθατε εδώ. Ελπίζω στην επόμενη συνεδρίαση να ακούσουμε καλύτερα νέα για τον κανονισμό αυτό. Ευχαριστώ την Κομισιόν, ευχαριστώ όλους σας όλους όσους έμειναν μέχρι το τέλος πιστοί. Αύριο έχουμε τους συντονιστές από ε, στις 9 και στις 10 και μισή έχουμε α, τη συνεδρίαση. Έρχεται και ο Υπουργός των Φαρόε. Το λέω για όσους ενδιαφέρονται. η υπουργό της της Ισλανδίας αποφάσισε να αρνηθεί την πρόσκλησή μας. Δεν θέλω να πω καμία κακία. Τι να πω, ας σταματήσουμε καλύτερα εδώ. στο εδώ λοιπόν και τα ξαναλέμε αύριο στις 9.